Okay. Λοιπόν, μπορούμε να ξεκινήσουμε. Καλησπέρα σε όλους. Ε, καλώς ήρθατε στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών και Νομισματικών Θεμάτων. Εάν δεν υπάρχουν ενστάσεις, θεωρώ ότι εγκρίνεται η μερίσια διάταξη. Δεν έχω κάποια ανακοίνωση αυτή τη στιγμή, επομένως μπορούμε να περάσουμε απευθείας στην ανταλλαγή απόψεων με τη Μαργρέτη Βερστάγκερ, εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρώπης ε, κατάλληλη για την ψηφιακή εποχή και για την απάντηση στην ε, πανδημία του κορονοϊού, του COVID-19. Ε, να καλωσορίσω λοιπόν την εκτελεστική αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και να την ευχαριστήσω για τη δυνατότητα που μας δίνει να συζητήσουμε για πρώτη φορά, να συζητήσουμε ε, το ρόλο της ε, βοήθειας ε, ως οικονομική απάντηση στην κρίση για τον ε, COVID-19 μετά από την πανδημία. Από την αρχή της κρίσης ήταν σαφές ότι χρειάζεται μία άνευ προηγουμένου οικονομική απάντηση για να αποφύγουμε την κατάρρευση του παραγωγικού μας συστήματα και σε μεγάλο βαθμό είδαμε ότι το σύστημα έκλεισε ε, λόγω του κορονοϊού. Ε, τα μέτρα τα οποία ελήφθησαν σε ευρωπαϊκό επίπεδο με την παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και το τέλος το πρόγραμμα ε, Ευρωπαϊκής, του Ταμείου Ευρωπαϊκής Ανάκτησης και Διάσωσης υπάρχουν δυνατότητε να υπάρχουν μέτρα για να ε, υποστηρίξουν τις οικονομίες με ένα προσωρινό πλαίσιο για να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα όσα προβλέπονται βάσει των κρατικών κανόνων. Μέτρα όπως ε, άμεσες ενισχύσεις, ε, επιλεκτικά φορολογικά κίνητρα, εγγυήσεις για δανειοδότηση επιχειρήσεων και ε, επιδοτούμενα ε, δάνεια, καθώς επίσης και γραμμές πίστοσες, οι οποίες θα επιτρέψουν στα κράτη-μέλη να δώσουν μια έγκαιρη και άμεση ε, απάντηση στις απειλές και να αποτελήσει και μια δυνατότητα, ένα μαξιλάρι που θα απορροφήσει την αρχική, τον αρχικό αντίκτυπο. κρίθηκε ένα πρώτο σύνολο τροπολογιών στο προσωρινό πλαίσιο που έδωσε επέκταση μέχρι και 800.000 ευρώ να επιχειρήσει 0% επιτόκιο και εγγυήσει ε, έως και 100% του κινδύνου και δυνατότητες ε, να δίνονται μέτρα ως κίνητρα για να υποστηρίξουν επιχειρήσεις που αναπτύσσουν και παράγουν προϊόντα για την καταπολέμηση του κορονοϊού όπως για παράδειγμα εμβόλια, φάρμακα, ε, ιατροτεχνολογικά προϊόντα και ούτω καθεξής. Και τέλος στις 8 Μαΐου είχαμε μια ακόμα σειρά τροπολογιών η οποία εγκρίθηκε ε, για ενίσχυση ε, για ανακεφαλαίωση ε, του χρέους, ανακεφαλαιοποίηση του χρέους ως ίστατη λύση. Όλα αυτά γίνονται σε στενή συνεργασία με τα κράτη-μέλη και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε περίπου 2-3 ευρώ σε κρατικές, κρατικές ενισχύσεις. Αλλά υπάρχει και μία ακόμα πτυχή την οποία πρέπει να λάβουμε υπόψη. Το τι μπορούν να κάνουν τα κράτη-μέλη προκειμένου να υποστηρίξουν τα παραγωγικό του συστήματο ε, και ε, αυτό σημαίνει ότι δεν είναι το ίδιο για κάθε ε, κράτος μέλος και φυσικά υπάρχουν διαφορετικές ανάγκες και δεν συνάδουν και με το μερίδιο του στην ευρωπαϊκή οικονομία. Το γεγονό λοιπόν ότι δεν έχουμε καθόλου ισότιμου όρου ανταγωνισμού και το γεγονό ότι υπάρχει και άνηση ε, αύξηση των φραγμών ε, και περαιτέρω κατακαιρματισμού είναι ε, κάτι το οποίο μας ανησυχεί ιδιαίτερα όσον αφορά την αγαστή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς και την βιωσιμότητα αυτών των μέτρων μεσοπρόθεσμα. Επομένως, η σημερινή συνεδρίαση πραγματικά αποτελεί μια πολύ σημαντική ευκαιρία για να γίνει μια ανταλλαγή απόψεων ε, για τον αντίκτυπο της κρατικής ενίσχυσης στην εσωτερική αγορά, στις οικονομίες των κρατών μελών και των οικονομιών, ε, όλων των διαφόρων οικονομικών τομέων και φυσικά και ε, ως προς το τι μέλη γενέστε στο εγγύς μέλλον. Χαίρομαι ιδιαίτερα λοιπόν που έχουμε εδώ τη Μαργκρέτε Βεστάγκερ μαζί μας, ώστε να μπορέσουμε να της απευθύνουμε όλα αυτά τα ερωτήματα. Πριν δώσω το λόγο στην Αντιπρόεδρο, επιτρέψτε μου να σας πω λίγο ε, πώς θα λειτουργήσει το σύστημα. Θα δώσουμε ε, πέντε λεπτά στην εκτελεστική αντιπρόσωπο για την εισαγωγική ε, παρέμβασή της και θα έχουμε ερωτήσεις και απαντήσεις. 10 ε, ερωτούντες, πέντε λεπτά, 2 λεπτά μέγιστο για την ερώτηση και τρία λεπτά για την απάντηση και αν επιτρέπετε μπορούμε, μας επιτρέψει ο χρόνος δηλαδή, μπορούμε να έχουμε και μια διαδικασία κάτσε στο τέλος. Να δώσω λοιπόν αμέσως το λόγο στην κυρία Βεστάγκερ. Έχετε το λόγο. Uh, Κυρία Βιστάγκερ, μπορείτε σας παρακαλώ να πατήσετε το κουμπί σας για να σας ακούμε. Ωραία. Τώρα. Τέλεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και σε ευχαριστώ Ειρήνη, για τα εισαγωγικά σου λόγια. Νομίζω ότι το τι έχει γίνει μέχρι Εκτιμώ ιδιαίτερα και ειδικά αυτή την εδώ το γεγονός ότι έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε τον διάλογό μας γιατί είναι ζητήματα τα οποία είναι πάρα πολύ σημαντικά και θα έχουν αντίκτυπο στους πολίτες ε, σε ολόκληρη την Ένωση. Η πανδημία αυτή έχει προκαλέσει πολλές ε, αλλαγές και πολλά βάσανα σε όλα τα κράτη-μέλη Άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, οικογένειες έχουν χάσει συγγενείς και ταυτόχρονα και η καραντίνα έχει σημαντικότατες κοινωνικές επιπτώσεις για τους ανθρώπους. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτή τη στιγμή να μην χάσουμε από τον προσανατολισμό μας το παρόν και ταυτόχρονα ανα, και ανανεώνοντας τις οικονομίες μας και τις κοινωνίες μας τις επόμενες εβδομάδες και μήνες με την προοπτική βεβαίως της πράσινης μετάβασης αλλά και της ψηφιακής μετάβασης. Την Τετάρτη η Επιτροπή θα παρουσιάσει πρόταση για ένα πακέτο ανάκαμψης. Η πρόεδρος Ursula von der έχει ήδη περιγράψει την αρχιτεκτονική αυτού του πακέτου εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στην τελευταία Ολομέλεια. Και τώρα οριστικοποιούμε το πακέτο αυτό, ώστε να μπορέσουμε να σας το παρουσιάσουμε μεθαύριο. Και χρειάζεται ένα τέτοιο σχέδιο ευρωπαϊκής ανά... που θα είναι ψηφιακό και πράσινο, ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επιδιώκουμε τους στρατηγικούς μας στόχους. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίως θα διαδραματίσει ουσιώδη ρόλο σε όλα αυτά διότι είναι σημαντικό το πακέτο αυτό να αποβεί σε όφελος όλων των Ευρωπαίων. Το Ευρωκοινοβούλιο θα έχει ίση συμμετοχή στη συζήτηση για το πώς θα επενδυθούν τα χρήματα, όπως και συμβαίνει με, την, το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ένα από τα ζητήματα που θέλω να σας θίξω σήμερα είναι το, ο νέος μηχανισμός ε, εξυγίανσης για εταιρείε που κατά τα άλλα είναι υγιείς, υγιείς όμως ε, έχουν αντιμετωπίσει κινδύνους λόγω της καραντίνας. Και βεβαίως θα επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα για να το συζητήσουμε ως προς τις λεπτομέρειες τους. Άπαξ και το παρουσιάσουμε συνολικά το πακέτο την Τετάρτη, όπως είπα. Όπως έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να κρατήσουμε ότι ορισμένα από τα βασικά μας στοιχεία θα μας βοηθήσουν σε αυτή την ανάπτυξη, ανάκαμψη που επιδιώκουμε. Η ενιαία αγορά προφανώς είναι ο βασικότερος παράγοντας για την ανάπτυξη, την απασχόληση και την ανταγωνιστικότητα. Ε, και η κρίση του κορονοϊού επιβεβαίωσε το πόσο σημαντικό είναι να διατηρηθεί αυτή η ενιαία αγορά. Οι κανόνες βεβαίως για την ενιαία αγορά συνεχίζουν να ισχύουν, γιατί η ενιαία αγορά θα αποτελέσει το βασικό κινητήρα και της ανάκαμψης, γιατί η ευημερία μας προέρχεται ακριβώς από το γεγονός ότι έχουμε εμπορικές συναλλαγές και ότι βρισκόμαστε σε σχέσεις αλληλεξάρτησης μεταξύ χωρών και πολιτών. Το σημαντικό στοιχείο λοιπόν είναι βεβαίως ότι αυτά θα συμβούν μόνο αν υπάρξει μια ενιαία αγορά χωρίς κατακαιρματισμούς. Άρα θα πρέπει να επιβάλλουμε και να ενισχύσουμε τους κανόνες που εσείς έχετε θεσπίσει ως νομοθέτες προκειμένου να εξασφαλίσουμε ότι η ενιαία αγορά δεν θα πληγεί από κατακαιρματισμό. Και γι' αυτόν τον λόγο εργαζόμαστε για να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της οικονομίας μας ιδίως ε, ε, ασκώντα κριτική και σε ορισμένα προστατευτικά μέτρα που έχουν ε, ληφθεί σε κάποια κράτη-μέλη. Η σχετική task force που έχει συσταθεί, έχει ήδη ε, συνεδριάσει και αυτό που είναι πολύ σημαντικό για εμάς να εξασφαλίσουμε είναι η λειτουργία της ενιαία αγορά. Για, τις, ε, για κανόνες κρατικών ενισχύσεων, στους οποίους αναφέρθηκε και η Πρόεδρος, βεβαίως αυτοί έχουν πολύ σημαντικό ρόλο στην ενίσχυση επιχειρήσεων σε αυτήν την άνευ προηγουμένου κρίση που αντιμετωπίζουμε. Έχουμε συνεργαστεί πολύ στενά με τα κράτη-μέλη προκειμένου να εγκρίνουμε 175 εθνικά μέτρα μέχρι σήμερα. Από τις αρχές Μαρτίου έως και σήμερα, επαναλαμβάνω, 175 τέτοιες αποφάσεις έχουν ληφθεί. Όπως είπα, όπως υπόθηκε μάλλον, προσαρμόσαμε τον ε, Μάρτιο και το προσωρινό πλαίσιο, κάτι που δίνει στην, τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη να έχουν την πλήρη προβλεπόμενη ευελιξία, ώστε να παρέχουν ρευστότητα και υποστήριξη προς τις οικονομίες τους. Το προσωρινό αυτό πλαίσιο έχει μάλιστα τροποποιηθεί δύο φορές έκτοτε, αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη των αναγκών των επιχειρήσεων. Συνολικά εξασφαλίζει ότι η κρατική ενίσχυση θα έχει περιορισμένο χρονικό χαρακτήρα και θα έχει στόχευση μόνο τα προβλήματα που πράγματι προκύπτουν από την κρίση του κορονοϊού η ε, υποστήριξη ρευστότητα μπορεί να παρασχεθεί έως και το τέλος, του, το τέλος του 2020 προκειμένου να μπορέσουν να αποφευθούν απολύσει, για να μπορέσει να συνεχιστεί η έρευνα, η ανάπτυξη, η ε, ε, έρευνα σε προϊόντα για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως το προσωρινό αυτό πλαίσιο επίσης διευκολύνει και την υποστήριξη ρευστότητας μέσω του χρέους. Καθώς εξελίσσεται η κρίση, πολλές, ε, πολλές επιχειρήσεις θα χρειαστούν κεφάλαια για να διατηρηθούν στη ζωή. Αν τα κράτη-μέλη θέλουν να, δίνουν τέτοια, να δώσουν τέτοια ενίσχυση, το πλαίσιο αυτό το προσωρινό εξασφαλίζει ότι θα υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι και περιορισμοί οι οποίοι θα αποκλείουν μπόνους και άλλα τέτοια μέτρα ώστε πραγματικά τα χρήματα να αξιοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο δίνονται. Και όταν χρησιμοποιούνται βεβαίως και αξιοποιούνται χρήματα των φορολογουμένων χρειάζεται διαφάνεια. Γι' αυτό και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να είναι πλήρως διαφανή για το πώς δόθηκαν οι κρατικές ενισχύσεις και πώς τα μέτρα που έχουν θεσπίσει πράγματι βοηθούν την εξυπηρέτηση του στόχου της ψηφιακής και πράσινης μετάβασης. Μέχρι στιγμής τα χρήματα που έχουν δοθεί από τα κράτη-μέλη μέσω τέτοιων ε, προγραμμάτων και σχεδίων ανέρχονται σε 2-3 εκατομμύρια ευρώ, ένα αδιανόητο, ε, αδιανόητα υψηλό ποσό βεβαίως. Ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλέ μεγάλες διαφορές μεταξύ των κρατών μελών και αυτέ αυτές οι διαφορές δεν αντικατοπτρίζουν μόνο την αλλαγή του μεγέθου των ε, κρατών μελών αλλά και των ε, διαφόρων βοηθειών και καθεστώτων υποστήριξης που παρέχονται σε, κάποια, σε όλα τα κράτη-μέλη. Και θα πρέπει κα, κανείς να την έχει αυτή τη διάσταση υπόψη του. Και γι' αυτόν τον λόγο, εν ώψη και στο πλαίσιο μάλλον του πολιτού δημοσιονομικού πλησίου και του μηχανισμού εξυγίανσης θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτή η κρίση δεν θα είναι μια, ένα ασύμετρο σοκ ε, εις βάρος των κρατών μελών, αλλά ότι θα είναι απλά ε, ένας, ένας μηχανισμός για να υποστηριχθούν επιχειρήσεις, να μην χαθεί η συνοχή που έχει επιτευχθεί με πολύ κόπο τα τελευταία χρόνια. Επίσης, Υπάρχουν ε, και ορισμένες επιπτώσεις της κρίσης του κορονοϊού όσον αφορά τον έλεγχο του ανταγωνισμού. Βεβαίως η κρίση αυτή έχει ε, προκαλέσει κάποιες ε, ελλείψεις όσον αφορά αναγκαίο υλικό για την αντιμετώπιση της πανδημίας, κάτι που οδήγησε και πολλές χώρες και επιχειρήσεις να προβούν σε συνεργασία. Οι κανόνες κατά των μονοπωλίων ε, βεβαίως δεν θα πρέπει να ε, εμποδίσουν τέτοιες μορφές συνεργασίας σε αυτή τη φάση τη ε, κρίση του κορονοϊού. Αυτό βεβαίω να το, ξε, το ξεκαθαρίσω ότι δεν σημαίνει ότι οι επιχειρήσει μπορούν να εκμεταλλευτούν την κρίση αυτή για να προχωρήσουν σε κατάχρηση τη δεσπόζουσα θέση του ή άλλε τέτοιε πρακτικέ. Στι 8 Απριλίου λοιπόν η Κομισιόν ενέκρινε προσωρινό πλαίσιο για την εκτίμηση των επιπτώσεων τη κρίση και στη σχετική ανακοίνωση μάλιστα αναφέρονται και συγκεκριμένα κριτήρια για το πώς μπορούν να υπάρξουν τέτοιες συνεργασίες. Επίσης προβλέπεται εκεί η δυνατότητα ε, έκδοσης συγκεκριμένων επιστολών έγκρισης κάποιων τέτοιων project συνεργασίας στη βάση πάντοτε αυτών των κανόνων. Και μια τέτοια επιστολή μάλιστα εγκρίθηκε και δημοσιεύθηκε και την ίδια μέρα. Αφορούσε τη συνεργασία μεταξύ φαρμακοβιομηχανιών για την αντιμετώπιση ελλείψεων κρίσιμου νοσοκομιακού υλικού και φαρμάκων για την θεραπεία των ασθενών του COVID-19 και όλα αυτά συνέβησαν στην, ε, με βάση τους κανόνες που ισχύουν ε, και με τα όσα είχαμε προβλέψει. Σχετικά με τον έλεγχο των συγχωνεύσεων, συνεχίζουμε να λαμβάνουμε αιτήσει και επεξεργαζόμαστε τις σχετικές αιτήσει ως συνήθως για να εξασφαλίσουμε μια ομαλή διαδικασία ε, υπό τις νέες αυτές ε, μορφές εργασίας εξ αποστάσεως και στο Κοινοβούλιο και στην ε, Κομισιόν και βεβαίως με πάντοτε, με σεβασμό των προθεσμιών. Η Κομισιόν έχει εκδώσει και κατευθυντήρες γραμμές για το πώς μπορεί κανείς να κοινοποιεί τέτοιες προτινόμενες συναλλαγές. Οι προκλήσεις που σχετίζονται με την εκτίμηση και την αξιολόγηση αυτών των ερευνών για, τους, ε, για τις συγχωνεύσεις είναι βεβαίως πολλαπλάσιες από ό,τι είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν πριν την κρίση, όμως εξακολουθούμε να ελέγχουμε κάθε περίπτωση ξεχωριστά, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ιδιαιτερότητες του κάθε κλάδου. Να ολοκληρώσω λέγοντας, λέγοντας ότι η δουλειά μας συνεχίζεται με πρωτοφανή ένταση Ξέρετε ότι η Στεφανή Γιονκοτών έχει υποβάλει, έχει παρουσιάσει και μια στρατηγική μας για την ανταγωνιστικότητα στην την ε, Ολομέλεια του Μαρτίου. Βεβαίως η κρίση άλλαξε τα σχέδιά μας, όμως θα έχουμε σύντομα ξανά την ευκαιρία να σας ε, ενημερώσουμε για την ε, για, τη για τα σχετικά μας σχέδια. Αποδείχθηκε ότι το Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για αυτόν τον τομέα πολιτική, ακριβώ γιατί είναι ένα τομέα πολιτική πάρα πολύ σημαντικό για την οικονομία μα. Και αυτό ισχύει τώρα περισσότερο από κάθε άλλη φορά. Παρά το ότι κάναμε κάποιε αλλαγέ στον τρόπο εργασία μα, δημιουργώντα ε, αυτά τα προσωρινά πλαίσια, δεν έχουμε σκοπό και δεν το έχουμε κάνει μέχρι στιγμή να αναστείλουμε την ισχύ των κανόνων ανταγωνισμού. Του χρειαζόμαστε αυτού του κανόνε και χρειαζόμαστε εντατική επιβολή των κανόνων αυτών ακριβώς για να ενισχύσουμε τις οικονομίες μας, να δώσουμε κίνητρα για την ανάπτυξη και την καινοτομία. Αυτά και άλλα πολλά θέματα βεβαίως πολύ ενδιαφέροντα θέλω να σήμερα να συζητήσω μαζί σας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, κύριε Αντιπρόεδρε. Να ξεκινήσουμε τώρα με τις ερωτήσεις. Να ξεκινήσουμε με τον κύριο Νίντερ Μάγερ από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, και καλώς ήρθατε, Επίτροπε. Ως συνήθως, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσω για την τόσο ε, κοπιώδη δουλειά σας τους τελευταίους μήνες. Τη δική σας και των συνεργατών σας. Βεβαίως, οι συνθήκες που αντιμετωπίζουμε είναι πρωτόγνωρες. Πρέπει λοιπόν να προχωρήσουμε γοργά. Τώρα ολοκληρώνεται η πρώτη φάση προκειμένου να υπάρξει ρευστότητα προς την αγορά. Δεν είχαμε χρόνο να σκεφτούμε όλες τις επιπτώσεις και το τι θα ακολουθήσει αλλά πρέπει να το κάνουμε ε, αμέσως. Γι' αυτό θέλω να επαναλάβω την ερώτηση της Προέδρου μας, της Ιρένε, και κάτι που το αναφέρατε κι εσείς. Μιλάμε εδώ για τις επιπτώσεις στήριξη στην οικονομία σε διαφορετικού βαθμού και στήριξη προ τι εταιρείε σε διαφορετικού βαθμού στα διάφορα κράτη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Από του αριθμού που μα δώσατε, βλέπουμε να υπάρχουν μεγάλε διαφορέ και αυτό στην πράξη θα έχει και διαφορετικό δημοσιονομικό αντίκτυπο. Αναφέρατε ότι το πολιτέ δημοσιονομικό πρόβλημα θα πρέπει να καλύψει και αυτά τα προβλήματα για να βεβαιωθούμε ότι η κρίση αυτή δεν θα αλλάξει εντελώ την σύσταση των εταιριών και το πώς ε, διαμορφώνονται τα μερίδια ιδιοκτησία τους. Θα πρέπει λοιπόν να μα πείτε από ε, τι αρμοδιότητέ σα τι μέτρα προτείνετε. Επίση, μια από τι βασικέ προτεραιότητε τη Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Επιτροπή την ε, αύξηση τη νομιμοποίηση και τη αυτοκυριαρχία τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, τις επάρκειες, ώστε να καλύψουμε και τις χώρες που είναι ε, πιο μακριά από το κέντρο και έχουν διαφορετικό οικονομικό μοντέλο. Είναι μεγάλη προτεραιότητα και για μας να είμαστε έτοιμοι για τις μελλοντικέ προκλήσεις. Διερωτώ με ωστόσο, πώς θα βεβαιωθούμε ότι οι προτεραιότητες αυτές θα μπορούν να συνδυαστούν με τη στήριξη προς τον ε, ανταγωνισμό για τις αγορές και την διαφάνεια, τη διαφάνεια των οικονομικών πολιτικών. Επίσης, πώς όλα αυτά θα μπορούν να είναι συνεπή με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική μας για τη στήριξη του δίκαιου και αμοιβαίους εποφελούς εμπορίου στον κόσμο. Σας ευχαριστώ κατά πρώτα για τις ευχαριστίες, για την ταχύτητα και την ποιότητα της δουλειάς μας. Θα τα μεταφέρω στους συνεργάτες μου. Εργάζονταν νυχθημερών, Επτά ημέρε την εβδομάδα. Κάποιε φορέ δεν κοιμόντουσαν κιόλα για να βεβαιωθούν ότι όλα θα προχωρήσουν όσο το δυνατόν ταχύτερα. Ευχαριστώ που το καταλαβαίνετε. Κατά δεύτερον, τις συνηθισμένες ημέρες βεβαίως υπάρχουν διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Εάν θέλουν να αξιοποιήσουν την ευελιξία που υπάρχει στους κανόνες για την κρατική βοήθεια, Λόγω χάρη δεν έχουν όλα τα κράτη-μέλη τέτοιο μηχανισμό για τις αγορές ηλεκτρικού ρεύματος ή ε, δεν μπορούν όλα να στηρίξουν τους χρήστες ε, που κάνουν χρήση εντατική ενέργειας. Αλλά οι διαφορές είναι πολύ μικρότερες από αυτό που βλέπουμε σήμερα στην πραγματικότητα. Δηλαδή, όταν περάσουμε στην επόμενη φάση, δεν θα είναι το πρόβλημα τόσο πολύ ρευστότητα, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό τα κεφάλαια. Τα κεφάλαια που χρειάζονται εταιρείε. Και αυτά θα υπόκειται σε διαφορετικέ προποθέσει. Διότι και εντό και μεταξύ κρατών μελών δεν μπορούν όλες οι επιχειρήσεις να έχουν την ίδια ε, προσφορά κεφαλαίου και πρέπει βεβαίω να σκεφτούμε ότι θα πρέπει να μειχθούν όσοι έχουν πληρώσει κανονικά του φόρου του, αλλά επίση να υπάρξουν και κίνητρα για τα κράτη ώστε να αναλάβουν πρωτοβουλίε και πάλι και οι επιχειρήσει να καταφέρουν να σταθούν και στα πόδια του και να είναι ανταγωνιστικέ. Και έπειτα, αν δοθούν κεφάλαια ε, σε ανταγωνιστέ, εάν κάποια εταιρεία είναι μεγάλη, α πούμε, θα πρέπει να δει πώ να αντισταθμίσει τι ενδεχόμενε τρευλώσει ανταγωνισμού σε μια δεδομένη αγορά, διότι θα υπάρξουν ανταγωνιστές που δεν πήραν τα ίδια κεφάλαια. Νομίζω λοιπόν ότι το αρχιτεκτόνημα της ανάκαμψης θα είναι πολύ σημαντικό και ως προς το εργαλείο της στήριξης στην ε, ε, πιστοτική ε, δυνατότητα και Στι βοήθειε που θα δοθούν, ώστε τα κράτη-μέλη να έχουν ένα σχέδιο για τι προσεγγίσεις του και τη στήριξη που θα δοθεί και να είναι βέβαια ότι θα προστατεύσουν την αλυσίδα παραγωγή αξιο... αγαθών και αξιών. Επίση, για το θέμα τη επικυριαρχία, ένα από τα πιο δυνηρά που ζήσαμε ήταν ότι είδαμε τομεί όπου υπήρχε εξάρτηση, ε, παρακεταμόλη, α πούμε, εξάρτησή μα από την Ινδία. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να διαφοροποιήσουμε την παραγωγή μα, αλλά ότι θα το σχεδιάσουμε αυτός μια αυτονομία στρατηγικού χαρακτήρα και αρκετά ανοιχτή δηλαδή ελεύθεροι. Να σκεφτούμε δηλαδή τι είδου ε, κινήσει θέλουμε να κάνουμε, τι μέγεθο να έχει η οικονομία μα, να μην ξεχνάμε ότι είμαστε και το μεγαλύτερο σύνολο χωρών ε, με εμπορικέ ε, σχέσει και παγκοσμίω. Θα πρέπει λοιπόν να έχουμε σχέσει ανοιχτέ, ελεύθερε με το παγκόσμιο εμπόριο και τι δυνάμει του. Αυτέ τι συζητήσει θα μα αποσχολήσουν τι ερχόμενε εβδομάδε. Πρόεδρο, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα Κάρμεν από του Σοσιαλιστέ και Δημοκράτε. Mrs. Avram, Κύριε Αβραμ, μπορείτε να πατήσετε το κουμπί. Speak. Could you press the speak button, please, Mrs. Avram? Yes. Ναι. Με ακούτε τώρα? ναι. Και σας βλέπουμε και σας ακούμε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Κυρία Επιτροπέ, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας και χαίρομαι που σας ξαναβλέπω, ακόμα και διαδικτυακά. Έχω αρκετές ερωτήσεις, επομένως θα περάσω απευθεία στο προκείμενο. Όσον αφορά όλε αυτέ τι κρατικέ ενισχύσει που θα δοθούν σε επιχειρήσει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση, γνωρίζουμε ότι δεν μπορούν ε, όλα τα κράτη-μέλη να βοηθήσουν τι επιχειρήσει του με τον ίδιο τρόπο. Θεωρείτε ότι ακόμα και χωρί το μηχανισμό και χωρί ε, το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, εξακολουθεί να υπάρχει κίνδυνο να αυξηθούν οι αποκλήσει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση μακροπρόθεσμα. Και επίση θα ήθελα να ρωτήσω τι γίνεται με την πολύ σημαντική ε, έρευνα ε, κρατικών ενισχύσεων για περιπτώσεις κρατικών ενισχύσεων ε, φερόμενες ότι συνέβησαν πριν από τον κορονοϊό. Είναι σε εξέλιξη ή έχουν παγώσει. Επίσης, ξέρουμε ότι τα μέσα αυτά δεν αρκούν γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση θα χρειαστεί και νέους πόρους για τις νέες στρατηγικότητες. Πρέπει να βρεθούν ήδη οι πόροι. Ε, υπέρ μια πρότασης ε, ψηφιακή φορολόγηση μέχρι το τέλο του έτου. Θεωρείτε ότι είναι εφικτό, θεωρείτε ότι τα μέτρα και η κρίση αυτή ε, επιτάχυναν κάπω τις διαδικασίε θα πρέπει να είμαστε αυτάρκοι σε πολλοί τομεί. Αυτό καταδείχθηκε από αυτή την πανδημία. Θεωρείτε λοιπόν ότι θα μπορέσουμε να έχουμε στήριξη όπω έχουμε στήριξη στου γεωργού και στον κλάδο τη γεωργία για να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση πιο ανεξάρτητη. Και θα ήθελα να κάνω και μία ερώτηση για τον ανταγωνισμό. Υπάρχει μεγάλη συζήτηση τώρα για τι ε, εφαρμογέ ηχνηλάτηση ε, του COVID που ε, αναπτύσσονται από μεγάλε επιχειρήσει και τίθεται θέματα και προστασία τη ιδιωτικότητα αλλά και πώ κάποιε πολύ μεγάλε επιχειρήσει μπορούν να συλλέγουν τώρα ε, πολλά ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα των πολιτών και των καταναλωτών. Ελοχεύει ο κίνδυνο να περιοριστεί ο ανταγωνισμό ακόμα περισσότερο προ όφελο αυτών των γιγάντων. Ευχαριστώ πολύ για τι απαντήσει σα και προσβλέπω ε, και ε, στο να συναντηθούμε διαζώσει για την έκθεση για τον ανταγωνισμό, ελπίζω. Ευχαριστώ πολύ και παρομοίω και εγώ εργάζομαι εντατικά μέσω διαδικτύου, με το Webex, ε, με αυτή την τεχνολογία και πιστεύω ότι αποδεικνύει ότι υπάρχουν ωφέλη αλλά και ελλείψεις. Και φυσικά ε, και εγώ περιμένω να σας συναντήσω και διαζώσει. Όσον αφορά τώρα την πρώτη σας ερώτηση, τις μακροπρόθεσμες διαφορές, ένας από τους λόγους ε, για τους οποίους είμαστε πιο αυστηροί όσον αφορά τις ε, εισρωές κεφαλαίων είναι ακριβώς διότι Θέλουμε να μειώσουμε τον κίνδυνο μακροπρόθεσμης στρέβλωσης του ανταγωνισμού. Ιδάλλως ε, υπάρχει ένας κίνδυνος ο οποίος ε, θα είναι συνεχής ε, τρόπον τεινά. Βεβαίω δεν μπορούμε να δώσουμε έγκριση για ενίσχυση η οποία θα είναι υπερβολική. Πρέπει να είναι ανάλογη με τις ανάγκες του καθενός. Και θεωρώ ότι το τι κάνει ένα κράτο μέλο, επηρεάζει και το τι θα συμβεί σε ένα άλλο κράτο μέλο, διότι ε, μπορούμε να έχουμε και στήριξη στις προμήθειε, επομένως μπορούμε να σας προμηθεύουμε προϊόντα ή οι πελάτες να ζητούν τα προϊόντα σας, επομένως υπάρχει μια βοήθεια και από εκεί. Θεωρώ όμω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε και σε αυτό και στη συζήτηση για τα μέσα διάσωση τα οποία θα παρουσιάσουμε την Πέμπτη. Όσον αφορά τις ε, έρευνες σε εξέλιξη, είναι σε εξέλιξη ακόμα αυτή τη στιγμή. Ίσως έχουν καθυστερήσει λίγο, διότι όλοι ασχολούνται με αυτές τις βραχυπρόθεσμες βοήθειες, αλλά δεν έχουν αναβληθεί και σε καμία περίπτωση δεν θα σταματήσουν. Τώρα, όσον αφορά τους ίδιους πόρους, συμφωνώ ότι χρειαζόμαστε περισσότερους ε, ίδιους πόρους για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και αυτό φυσικά σε κάποιο βαθμό διαφέρει από τη συζήτηση για την ε, ψηφιακή φορολόγηση, διότι η ψηφιακή φορολόγηση είναι σημαντική ανεξάρτητα από το τι άποψη έχει κάποιος για τους ιδίους πόρους. Βλέπετε πώς ε, οι φορολογούμενοι υποστηρίζουν τις επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή και νομίζω ότι είναι κατεπήγον όχι μόνο οι περισσότερε επιχειρήσει να καταβάλουν του φόρου του, αλλά όλε οι επιχειρήσει να καταβάλουν του φόρου του. Εγώ ελπίζω να υπάρξει μια συνολική συνένεση από αυτού, αλλά σε περίπτωση που δεν υπάρξει, εξακολουθώ να θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό εμεί στην Ευρώπη να ε, υποβάλουμε μια πρόταση και να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υπάρχει συνένεση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Διότι θα πρέπει κάθε επιχείρηση να καταβάλει του φόρου τη όταν εργάζονται διαδικτυακά, όπω κάνουν και και ε, με τις υπόλοιπε δραστηριότητες. Ε, δίνεται πολύ μεγάλη στήριξη και νομίζω ότι αυτό που έχει πολύ μεγάλη σημασία εδώ είναι να αξιολογήσουμε τι αγορά θέλουμε να είμαστε. Αυτή η ιδέα μιας ανοιχτής στρατηγικής οικονομίας θα μπορούσε ίσως να ανοίξει το δρόμο. Ε, από μια θα έχουμε ε, μια νέα ανθεκτικότητα, θα είμαστε πιο καλά προετοιμασμένοι και θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα περισσότερο, διότι το τραπεζικό μας σύστημα είναι σε τελείως διαφορετική κατάσταση από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Επομένως μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, το να μπορούμε εμείς να διεξάγουμε τις δραστηριότητές μας όπως πρέπει, διότι βασιζόμαστε πολύ στο εμπόριο και δεν θα πρέπει να το χάσουμε αυτό στη διαδικασία μια προσπάθεια μεγαλύτερη ανθοκτικότητα και μεγαλύτερη αυτονομία. Τώρα, όσον αφορά τι εφαρμογέ συχνηλάτηση του COVID-19, νομίζω ότι και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη να δώσουν τη δυνατότητα στου πολίτε να έχουν τη δυνατότητα να ιχνηλατούν τον ιό. Όταν συνεργαζόμαστε με τους ε, γίγαντες σε ψηφιακό επίπεδο είναι για να μπορέσουμε να είμαστε ε, βέβαιοι ότι θα υπάρχει μια εφαρμογή στο σύστημά σας που θα λειτουργεί, πραγματικά θα ανοιχνεύει τον ιό και θα μπορείτε να χρησιμοποιείτε και διαφορετικές εφαρμογές για να γίνει αυτό και διασυνοριακά ε, και φυσικά με διαφορετικά λειτουργικά συστήματα στα τηλέφωνά σας. Και νομίζω ότι αυτό είναι αυτό που έχει τη μεγαλύτερη σημασία. Και τέλος, κατ' εξίσου σημαντικό, θα πρέπει οι πολίτες να νιώθουν ασφαλείς με τη χρήση της εφαρμογής. Αν εμπιστεύονται την τεχνολογία δεν θα το χρησιμοποιήσουν, δεν θα χρησιμοποιήσουν την εφαρμογή ε, και δεν θα την κατεβάσουν φυσικά. Ευχαριστώ. Ο Λουίς Καρικάνο τώρα από το Ρινιού. Um, Νομίζω με ακούτε, αλλά δεν μπορείτε να με δείτε. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπε, δεν ξέρω γιατί δεν λειτουργεί η κάμερά μου. It's the secretariat here, Mr. Garrick. Σας μιλάει η γραμματεία. Ναι, σας ακούμε, αλλά δυστυχώς πράγματι δεν μπορούμε να σας δούμε. Κύριε Γαρικάνο. Should I take... Θέλετε να περιμένω ένα λεπτό, γιατί νομίζω ότι οι διερμηνείς ε, δεν μπορούν να εργαστούν αν δεν με βλέπουν. Σωστά. Please continue with the question. Συνεχίστε με την ερώτηση σας παρακαλώ. Now it's good. Thank you. You, you... Α, ωραία. που αντιμετωπίζουν κινδύνους λόγω του κορονοϊού. Ε, θέλω να σας ρωτήσω σχετικά με τον σχεδιασμό και την αρχιτεκτονική αυτού του μηχανισμού, γιατί χρειαζόμαστε και τις γνώσεις, όμως χρειαζόμαστε και τη διαθεσιμότητα να μπορέσουμε να παρακολουθήσουμε την εφαρμογή ενός τέτοιου μηχανισμού. Ακριβώς γιατί δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη πείρα. Θέλω να μου πείτε την άποψή σας για, τα τρία σενάρια. Ότι η θα έχει τη βασική εντολή. Εγώ προσωπικά νομίζω ότι δεν μπορεί κάτι τέτοιο να γίνει μέσω των εθνικών δηλαδή τραπεζών μετά. Δεύτερο είναι να ζητηθεί από τα κράτη-μέλη να δημιουργήσουν ε, ταμεία για τη διάθεση αυτών των χρημάτων, κάτι που επίσης με βρίσκει αντίθετο γιατί είναι ευρωπαϊκά χρήματα αυτά. Η τρίτη πιθανότητα, δυνατότητα λοιπόν είναι να δημιουργηθεί ένα ε, ένας μηχανισμός ο οποίος θα ε, συγχωνεύει κρατικούς και ιδιωτικούς επενδυτές μέσω της ε, μορφής των ε, συμπράξεων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα και ότι η Κομισιόν θα εγγυάται την κεφαλαιακή επάρκεια έως και ένα επίπεδο 11%. Ε, συμφωνείτε με μια τέτοια προοπτική ή εσείς θα προτιμούσατε μια διαφορετική δομή, μια διαφορετική αρχιτεκτονική. Σας ευχαριστώ πολύ και προσβλέπω βεβαίως και στην ε, παρουσίαση που θα κάνει η Κομισιόν την Τετάρτη νομίζω ότι θα είναι πολύ φιλόδοξη. Θα ευθυγραμμίζεται και με την γαλλογερμανική πρόταση που κατατέθηκε τις προηγούμενες εβδομάδες και νομίζω ότι θα δώσει και τη σωστή απάντηση στις προκλήσεις, όσον αφορά τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι οικονομίες Η κυρία Βεστάγκη, σας ευχαριστώ. Δεν έχουμε ακόμη ξεκινήσει, η αλήθεια είναι, την εφαρμογή αυτού του μηχανισμού. Τώρα οριστικοποιούμε κάποιες τελευταίες λεπτομέρειες και να σας πω την αλήθεια, δεν νομίζω ότι θα ε, μπορούσα να σας πω το οτιδήποτε προτού μπήκε η τελευταία ε, πινελιά από το Κολέγιο των Επιτρόπων. Την Τετάρτη λοιπόν. Ένα όμως ε, που κρατώ από αυτά που είπατε και που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, όλα όσα είπατε βεβαίως είναι σημαντικά, αλλά υπάρχει ένα θέμα το οποίο θέλω να αναδείξω. Και αυτό είναι ότι αυτό που είπατε ότι ε, ε, η, τα, τα κεφάλαια αυτά θα πρέπει να είναι καινούρια. Και βεβαίως χρειάζεται εμπειρογνωμοσύνη για να μπορέσουν να αξιοποιηθούν γρήγορα και αποτελεσματικά. Και βεβαίως εγώ θα ε, εξασφαλίσω στο μέτρο των δυνατοτήτων μου ότι αυτές, αυτοί οι κανόνες θα ισχύσουν και ότι σε αυτήν την κατεύθυνση θα κινηθούμε. Ξέρετε, πολλές φορές λένε ότι δικαιοσύνη που απονέμεται αργά δεν είναι δικαιοσύνη. Έτσι και με αυτά τα χρήματα. Αν φτάσουν αργά, τότε θα είναι άχρηστα πλέον σε εκείνους που τα χρειάζονται. Και ένα από τα σημεία που έχω ε, παρατηρήσει εγώ σε σχέση με αυτή την πρόταση είναι οι διαφορέ ανάμεσα στα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη θέλαν πολύ αυτές τις ε, τράπεζε προώθηση, προώθησης, άλλα κράτη-μέλη έχουν νέε τράπεζε προώθηση ή μπορεί να μην έχουν ε, μεγάλη εμπειρία, κάποια άλλα κράτη-μέλη έχουν μεγάλη εμπειρία με τέτοιου είδους ταμεία, κάποια είναι άπειρα. Γι' αυτό και εγώ θέλω να συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα σε βάθος με εσάς και με τα κράτη-μέλη, ελπίζοντας ότι θα μπορέσουμε να βρούμε τρόπους ώστε να εξασφαλίσουμε ότι το εργαλείο αυτό, ο μηχανισμός αυτός, πράγματι στα κράτη-μέλη θα δώσει τη δυνατότητα να δώσουν στις επιχειρήσεις τους την φερικιότητα, τη ρευστότητα που δεν μπορούν να βρουν διαφορετικά. Και ελπίζω να εξασφαλίσουμε αυτή την ευελιξία γιατί η ευελιξία είναι σημαντικό ώστε ταχύτατα να δοθούν τα χρήματα αυτά στι επιχειρήσει εκεί που χρειάζονται και ώστε οι αλυσίδε αξία να μπορέσουν να υποστηριχθούν εκεί όπου υπάρχουν πραγματικέ ανάγκε. Με αυτά που είπατε εσείς λοιπόν και στη βάση των όσων είπατε εσείς, εγώ σας εγγυώμαι ότι προσβλέπω πάρα πολύ στο να εργαστούμε με αυτόν τον τρόπο. Ευχαριστούμε και τώρα ο κύριος Γκουιφό από τους Πρασίνους. Πρόεδρε, ε, ο κύριος Γκριφό δεν φαίνεται... Α, ε, ναι, είναι συνδεδεμένος. Με ακούτε? Καλησπέρα σα Επίτροπε. Θεωρείτε ότι πέρα τη στήριξη των ε, επιχειρήσεων που έχουν δυσκολίε, δεν θα πρέπει να δούμε τη βοήθεια και στην περίοδο μετά την κρίση, που θα πρέπει να ε, είναι μεγαλύτερο στην, ε, στις, επεξεργασία, επιχειρήσεις επεξεργασίας πράσινης και οικολογικής παραγωγή. παραγωγής. Εδώ έχουμε μια πράσινη ρεσιμότητα στην Ευρώπη για τις επιχειρήσεις με δυσκολίες. Και δεν συμφωνούν βεβαίως όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, αυτοκινητοβιομηχανία και πραγματικά βλέπουμε καθημερινά να υπάρχουν πολλές ε, επιδοτήσεις σε κλιματοκτόνες και επιχειρήσεις που δεν σέβονται τις, τα περιβαλλοντικά πρότυπα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ε, κατά πόσον μπορούν να συμβάλλουν όλα αυτά στους στόχους μας, ε, όπως και στο Πράσινο Σύμφωνο. Θα πρέπει να δούμε στην περίοδο μετά της κρίσης, εάν το status quo που θα δημιουργηθεί θα είναι επιζήμιο για τα είδη των ζώων του πλανήτη και για το περιβάλλον. Θα πρέπει να σκεφτούμε τις επιχειρήσεις που ρηπαίνουν και να δούμε εάν οι πράσινες επιχειρήσεις επιτρέπουν τις οικολογικές επενδύσεις ε, με κλιματικούς στόχους. Η ερώτησή μου λοιπόν αφορά το θέμα της έλλειψης πράσινης ερωσιμότητας για τις βοήθειες που θα δοθούν ε, μετά την κρίση. Και αυτό για λόγους ενδεχομένως πολιτικούς, δεν ξέρω. Και να ρωτήσω και το εξής αυτή τη στιγμή τι ε, οικολογικέ και κλιματικές ε, βλάβες κάποιων δραστηριοτήτων τι πληρώνουν οι περιφερειακές και δημοτικές αρχές. Και θα πρέπει να δούμε ε, το κλιματικό κόστος, ποιες επιχειρήσεις θα το αναλάβουν, αυτές που καταναλώνουν άρθρακα ή όχι, στα πλαίσια του Πράσινου Συμφώνου. Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Επίτροπε, πιέστε το κουμπί σα. Ναι, δεν ε, ήξερα αν έχει ολοκληρώσει την ερώτηση του Κλοντ. Ε, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία μας είχαν απασχολήσει ε, πολύ Και πρέπει να δούμε την πρόταση ανάκαμψης με το ε, δημοσιονομικό πλαίσιο και ξέρω ότι δεν υπάρχει έλλειψη πολιτικής βούλησης, αλλά εγώ το βρίσκω καθοριστική σημασίας. Αυτή η επιλογή μας, να πούμε ότι έχουμε έναν προπολογισμό για πολλά χρόνο, χρόνια, με ένα αρχιτεκτόνημα ανάκαμψης γύρω από αυτό. Και αυτό θα περάσει όχι μόνο από κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και θα έχει και όλε τι απαραίτητε προποθέσει για να αποφύγουμε κάθε είδο κακοδιαχείριση ή εσφαλμένη ε, χρήση. Και να είμαστε βέβαιοι ότι θα επιδέκονται στόχοι που έχουμε συμφωνήσει και για την οικολογική ταυτότητα τη Επίρου μα και για να αξιοποιήσουμε τα ψηφιακά εργαλεία. Βεβαίω σκεφτόμαστε πολύ προσεκτικά σε τι βαθμό θα μπορούν αυτά να ισχύσουν και για την κρατική βοήθεια. Πάντως το βασικό εδώ είναι η νομική βάση, η νομική βάση που θα χρησιμοποιήσουμε. Φυσικά οι συνθήκε τώρα είναι έκτακτε και τη νομική βάση μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε αναλόγως. Με ευελιξία στην κρατική βοήθεια. Όμω θα πρέπει να δούμε τι βοήθεια πρέπει να δώσουμε στι επιχειρήσει για να επιβιώσουν. Όχι να κάνουν κάτι καινούριο, όχι για να αποκτήσουν νέε δυνατότητε παραγωγή, κάτι που δεν μπορούσαν να κάνουν προηγουμένω μόνε του. Θα πρέπει να είναι εταιρείε υγιεί. Ούτω ή άλλω και βοήθεια να του επιτρέψει να μην βυθιστούν ε, λόγω του απαγορευτικού και του lockdown σε αυτέ τι έκτακτε περιστάσει. Αυτό βεβαίω ε, δημιουργεί την εξή δυσκολία το γεγονό ότι υπάρχει ακριβώ αυτή η βοήθεια επιτρέψει μια επιχείρηση να επιπλέψει και από πάνω η Επιτροπή δίνει και οδηγίε για την πράσινη κατεύθυνση. Έτσι, αποφασίσαμε να πούμε ότι αν τα κράτη-μέλη το θέλουν, μπορούν να το κάνουν αυτό, ε, θα το ενθαρρύνουμε οι δυνατόν, γιατί κάποιες φορές το να επιπλέψει κανείς είναι ευκολότερο να κάνει πράσινες επιλογές. Πάντως, τα κράτη-μέλη, χρησιμοποιώντα τα χρήματα των φορολογουμένων ε, εντό του ίδιου κράτου μέλου που φορολογήθηκαν οι πολίτε, μπορεί να φανεί τελικά και το όφελο για τους ίδιου. Βεβαίω, μιλάμε για κονδύλια ενό ευρωπαϊκού ε, αρχιτεκτονήματο. Πάντω, σα διαβεβαιώ ότι δεν είναι έλλειψη πολιτικής βούλησης. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε πολύ. Ο κύριος Φανόφερτ, θέλω από τους συντηρητικούς μεταρρυθμιστές. Ευχαριστώ κύριε Βεστάγκερ που είστε εδώ μαζί μας και να σας συγχαρώ πραγματικά για την εξαιρετική δουλειά που έχει γίνει σε αρκετούς τομείς της αρμοδιότητάς σας. Τρεις ερωτήσεις έχω. Πρώτον, φαίνεται να υπάρχει μία επιστολή του τομέα ψηλή τεχνολογία που ζητά περαιτέρω μέτρα για του ε, κανόνε για τι κριτικές ενισχύσει και φυσικά ζητούν περαιτέρω χαλάρωση σε κάποιε κατευθύνσει. Θα ήθελα ε, να μου απαντήσετε στο κατά πόσον σκοπεύετε να κάνετε κάτι τέτοιο και αν ναι, με ποιο τρόπο. Δεύτερον, είδαμε και το έχουν γράψει και αναλυτικότατα οι Financial Times. Ε, επιθέσεις ουσιαστικά κατά ευρωπαϊκών ε, μετοχών. Παρακολουθείτε κάτι τέτοιο ε, και ε, σκοπεύετε να λάβετε κάποια μέτρα για να αντιμετωπίσετε αυτή την μάλλον αρνητική εξέλιξη. Και η τρίτη μου ερώτηση είναι τι κάνουν οι μεγάλες διεθνείς επιχειρήσεις. Υπήρχε στο Bloomberg μία ανάρτηση για ε, κινέζικες επενδύσεις σε πιο ανθεκτικά ε, στοιχεία ενεργητικού όπως τα αποκαλούν. Εσείς αναφερθήκατε ήδη στην ανάγκη να προστατευτούμε εναντίον επιθετικών ε, κινέζικων εξαγορών. Ε, το περιορίζεται αυτό μόνο σε κινέζικους ομίλους ή και σε άλλες χώρες, για να μην μιλήσω για τις Ηνωμένε Πολιτείε. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και σας ευχαριστώ επίσης και για τη συγχαρητήριά σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για μένα, γιατί βλέπω πόσο μεγάλη προσπάθεια γίνεται και όπως γνωρίζετε και εσείς ε, πολύ καλά, όπως και οποιοδήποτε άλλος που εργάζεται με τέτοιες συνθήκες, είναι κάτι τελείως διαφορετικά να εργάζεται κάποιος όταν ο καθένας βρίσκεται σε ένα διαφορετικό σημείο. Και σας ευχαριστώ πολύ λοιπόν για τα συγχαρητήρια υπάρχει ένα πολύ σημαντικό θέμα υψηλής προτεραιότητας, ε, το οποίο είναι ε, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι ο τρόπος που θα ορίσουμε την υγιή επιχείρηση δεν θα αποκλείσει κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες ε, έχουν προγραμματισμένη οικονομική στάση που τις κάνει να φαίνονται ε, επιχειρήσεις οι οποίες αντιμετωπίζουν δυσκολίε, αλλά στην ουσία είναι υγιεί γιατί είναι καινοτόμε, επιχειρήσεις, έχουν επενδυτέ, έχουν υποστήριξη και σε σύγκριση όμως με αυτό το οποίο θα βλέπαμε σε μια πιο όρημη επιχείρηση που θα είχε κάποιους πιο συμβατικού κανόνες, δεν θα ε, μπορούσαμε να πούμε ότι εντάσσονται σε αυτό το πλαίσιο. Ε, αυτή τη στιγμή λοιπόν βρίσκουμε μεμονωμένες λύσεις ε, για την κάθε περίπτωση, αλλά θέλουμε να εξασφαλίσουμε αντί να λαμβάνονται μεμονωμένες αποφάσεις, να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο οριζόντια προσέγγιση, διότι είναι υπερβολικό. Κάποιες από αυτές τις επιχειρήσεις είναι και σχετικά μικρές επιχειρήσεις και επομένως είναι και πάρα πολύ σημαντικό για μας ε, οι ορισμοί μας να έχουν και ένα περιθώριο για να λάβουν υπόψη ε, ε, και τις διαφορές σε αυτή τη θέση, γιατί μια καινοτόμος επιχείρηση, μια νεοφυής επιχείρηση μπορεί να είναι πολύ υγιή στη δομή της, αλλά να έχει ένα προγραμματισμένο προφίλ ε, για το κεφάλαιο που εκ πρώτης ε, να την κάνει να μοιάζει ως μια επιχείρηση που δεν εντάσσεται σε καμία από τις κατηγορίες μας. Αυτό λοιπόν είναι απόλυτη προτεραιότητα. Πρέπει να επιληθεί όχι μόνο στις μεμονωμένες αποφάσεις, αλλά και γενικότερα δεν ε, παρακολουθώ το θέμα αυτό των ε, hedge funds, ε, θα το εξετάσω και αν υπάρξει κάποιο πρόβλημα, πολύ ευχαρίστως να σας απαντήσω και να επανέλθω με μια απάντηση. Ήμουν στην αρχική μου ακρόαση που έχει καιρό πλέον που έγινε, δεν αναφέρθηκα σε ποια περιοχή ε, του κόσμου θα πρέπει ε, να εξετάζουμε κάποια πράγματα με μεγαλύτερη επαγρύπνηση. Διότι υπάρχει ε, και το θέμα της διάσωσης και δεν διασώζεται κάθε περιοχή του κόσμου με τον ίδιο ρυθμό. Και πρέπει λοιπόν εδώ να επαγρυπνούμε. Σκοπεύουμε να παρουσιάσουμε μια λευκή βίβλο για ξένες επενδύσεις, για εξαγορές, από ξένες ε, κρατικές επιχειρήσεις ή από επιχειρήσεις οι οποίες υποστηρίζονται από το κράτος ε, σε άλλες χώρες και φυσικά θα πρέπει να δούμε και αυτή τη μορφή τους επενδυτές. Ναι, αφενός εμείς ε, είμαστε ανοιχτοί ως Ευρώπη, αλλά πρέπει να έχει κάποιες κατάλληλες προθέσεις. Αν όχι, υπάρχει πρόβλημα. Και φυσικά τμήμα του προβλήματος είναι ότι θα πρέπει να μπορέσουμε να αυξήσουμε και την αμοιβαιότητα, διότι ναι μεν εμείς ε, είμαστε ανοιχτοί και διαθέσιμοι, αλλά θα πρέπει και οι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις να είναι εξίσου ευπρόσδεκτες σε άλλα μέρη του κόσμου. Πρέπει λοιπόν του κόσμου να εντείνουμε τις εργασίες μας και να ε, εξετάσουμε λίγο ε, τι γίνεται με τους ξένους παράγοντες στην ευρωπαϊκή οικονομία και τι μπορούμε να κάνουμε από αυτό; Ευχαριστώ πολύ. Ο Μικ Γόλας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι κανόνες κρατικής ενισχύσεων, κρατικών ενισχύσεων ε, έχουν ως στόχο να μην υπάρχει κρατική παρέμβαση όσο το δυνατόν περισσότερο. Όμως αυτοί οι κανόνες βασίζονται στην εσφαλμένη παραδοχή ότι ο καπιταλισμός είναι δίκαιος και αυτορυθμίζεται. Όμως φαίνεται τελικά ότι ο νεοφιλελευθερισμός μπορεί να λειτουργήσει μόνο με κρατικές ενισχύσεις. Είπατε ότι έχετε εγκρίνει 1,9 τρισεκατομμύρια για εθνικά συστήματα ενίσχυσης που προβλέπονται. Και δεν κατάλαβα. Εσείς ε, συστήνετε να υπάρχει περιβαλλοντική εστίαση αυτών των σχημάτων, χωρίς να υπάρχει όμως σχετική υποχρέωση, σωστά. Για χρήματα των φορολογουμένων μιλάμε. Ενώ θα ήταν μια εξαιρετική ευκαιρία να εξασφαλίσετε ότι οι περιβαλλοντικές προϋποθέσεις θα ήταν ενταγμένες στη συμφωνία αυτή. Είπατε ότι τα χρήματα αυτά απλά θα διατηρήσουν στη ζωή της επιχειρήσης. Εγώ δεν, δεν ικανοποιούμαι με αυτή την απάντηση. Αυτό που έχουμε δει είναι ότι κάποιες χώρες έχουν εισαγάγει κάποιες προϋποθέσεις όπως η Γαλλία, ενώ άλλες χώρες δεν έχουν θέσει καμία προϋπόθεση για να παρθούν αυτά τα χρήματα. Άρα δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού. Εγώ θεωρώ ότι οι κανόνες ε, κρατικών ενισχύσεων θα έπρεπε να είναι συμβατοί με τη Συμφωνία των ε, Παρισίων. Και βλέπουμε χώρες όπως η Γερμανία με, με πολύ δυνατή ισχυρή θέση να δίνουν κρατικές ενισχύσεις. Ενώ στην Ιρλανδία οι κανόνε κρατικών ενισχύσεων είναι στην πραγματικότητα κανόνε λιτότητα, περιορισμού του πώ η βοήθεια μπορεί να δοθεί σε επιχειρήσει. Για παράδειγμα, μπορούμε να βοηθήσουμε τι μικρέ μα επιχειρήσει. Θα βοηθήσει η Κομισιόν σε μια τέτοια κατεύθυνση, σε αυτό το τομέα, διότι οι μικρέ επιχειρήσει χρειάζονται την ε, βοήθεια αυτή περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο για να μπορέσουν να επιβιώσουν στην κρίση. Διότι αν δεν υπάρξει βοήθεια προς τις μικρές επιχειρήσεις δεν θα καταφέρουν να επιβιώσουν. Είναι προετοιμασμένη η Κομισιόν να παρέμβει σε αυτόν τον τομέα, να εξασφαλίσει ότι τα κράτη-μέλη θα δώσουν βοήθεια στις μικρές τους επιχειρήσεις. Αναμφίβολα. Οι κανόνες κρατικών ενισχύσεων πολλές φορές μας έχουν απαγορεύσει ακόμη και το να φτιάξουμε εστίες, εργατικές για παράδειγμα, κατοικίε. Έπρεπε να το κάνουμε μέχρι ΣΔΙΤ. Δεν, έχουμε, δεν είχαμε πολλές φορές τα χρήματα. Κάτι που έχει οδηγήσει στην εφαρμογή των κανόνων αυτών τελικά να καταλήγουμε στην επιβολή της λιτότητας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Επίτροπος. Δεν έχω να προσθέσω κάτι όσον αφορά τις, τους, τις περιβαλλοντικές προϋποθέσεις για τις κρατικές ενισχύσεις. Να πω όμως μία σκέψη. Νομίζω ότι οι νεοφιλελεύθεροι θα ήταν πολύ απογοητευμένοι βλέποντας την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρατηρώντας το τι κάνει. Δεν νομίζω ότι ισχύουν αυτά που περιγράψατε. Αντιθέτως, εγώ νομίζω ότι υπάρχει, έχουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς στην Ευρώπη. Στο πέρασμα των δεκαετιών ρεαλιστικά αναγνωρίσαμε εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ο καπιταλισμός στην ακατέργαστη μορφή του δεν είναι κάτι που το θέλουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές ως δημόσιος τομέας καταλαμβάνει μεγάλο κομμάτι της οικονομίας των οικονομιών μας, όπως και θα έπρεπε κατά τη γνώμη μας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα πώς τα δημόσια οικονομικά θα κατευθύνονται με ένα τέτοιον τρόπο ώστε να ε, διευκολύνεται το εμπόριο, να μην στρεβλώνεται η αγορά, ώστε να μπορεί να υπάρχει μια ενιαία αγορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό είναι ακριβώς αυτό που έχω προσπαθήσει να ξεκαθαρίσω κι εγώ. Πότε μπορούν να, μπορούν να δίνονται κρατικές ενισχύσεις, πότε δεν μπορούν να δίνονται κρατικέ ε, ε, ενισχύσει, πότε μπορούν πρωτοβουλιακά να κινούνται τα κράτη-μέλη, πότε θα πρέπει να κοινοποιείται κάτι εκ των προτέρων στην Κομισιόν. Όλα αυτά. Αυτό που όμω είναι πολύ σημαντικό για εμένα είναι ότι οι αιρετοί βουλευτέ του Ευρωκοινοβουλίου και των Εθνικών Κοινοβουλίων θα έχουν την νομιμοποίηση να πλαισιώσουν τη βάση των όσων θα γίνουν. Μπορούμε να πούμε ότι δεν θα δεχτούμε παιδική εργασία, κακές ή επισφαλείς συνθήκες και όρους εργασίας. Δεν θα επιτρέψουμε να πούμε ότι εξαιτίας αυτής της κρίσης θα καταστρέψουμε τον ε, υδροφόρο ορίζοντά μας ή το περιβάλλον. Θέλουμε δηλαδή με άλλα λόγια μέσω των δημοκρατικών δυνάμεων, μέσω των δημοκρατικών διαδικασιών να πλαισιώνουμε, να θέτουμε το πλαίσιο αν θέλετε της λειτουργίας αγοράς. Και εκεί εκεί αφού πλέον θα έχουμε φτιάξει αυτό το πλαίσιο που θα αντικατοπτρίζει τις αξίες μας, τότε ναι θα μπορεί να λειτουργεί η αγορά στη βάση των ε, κανόνων που ισχύουν. Του τι μπορεί κανείς να παράγει, τι θέλουν οι πελάτες, τι θέλουν οι καταναλωτές. Νομίζω ότι η ευρωπαϊκή δημοκρατία είναι, πολύ, είναι κάτι πολύ ευρύτερο από έναν απλό καπιταλιστικό παράδεισο. Και το βλέπετε αυτό και σε, κράτη -μέλη, σε πολλά κράτη-μέλη όπου η ισότητα δεν είναι δεδομένη. Ε, όλα αυτά, βεβαίω, οι ανισότητε είναι πολύ μικρότερε από ό,τι σε άλλα μέρη του κόσμου. Βεβαίω, έχουμε πολλά ακόμη να κάνουμε. Υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωση. Εμεί προσπαθούμε τελικά να αξιοποιήσουμε τα ωφέλη του καπιταλισμού προκειμένου να διαμορφώσουμε μια κοινωνική οικονομία της αγοράς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Αντιπρόεδρε, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση σε σχέση με τα νησιά και την νησιωτικότητα, διότι για στην ε, όλη μεταρρύθμιση για τις κρατικές βοήθειες πολλά κράτη που έχουν νησιά και εγώ είμαι από την Ιταλία, την Ιταλία που έχει πολλά νησιά, μεταξύ των οποίων δύο από τα μεγαλύτερα νησιά της Μεσογείου, τη Σικελία και τη Σαρδινία. Τα κράτη λοιπόν αυτά ζητούν έντονα το άρθρο βάσει του άρθρου 154 τη συνθήκη Λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προβλέψει τη δυνατότητα να δημιουργηθούν στα νησιά τέτοια συνθήκες ανταγωνιστικότητα που θα επιτρέψει να επιβιώσουν, γιατί έχουν λιγότερο δυνατότητα να ανταγωνιστούν, ακριβώς λόγω της γεωγραφικής τους θέσης. Ε, οι λόγοι εδαφικής συνοχής υποχρεώνουν τα κρατημέλη βάσει των κανόνων ανταγωνιστικότητας και ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να σκεφτούν τι ακριβώς θα να κάνουν για τα νησιά με τις ανάλογες διασυνδέσεις και για τη μεταφορά εμπορευμάτων και για να μην υπάρχει αυτή η δομική ανισότητα ανταγωνιστικότητας που έχουν σε σχέση με τις περιοχές ε, της πρωτικής χώρας. Αυτά πολύ συχνά ε, διωγγώνονται σε μείζωνα προβλήματα. Στο μέλλον λοιπόν, στην αναθεώρηση των κρατικών βοηθειών που θα δοθούν σκέφτεστε να συμπεριλάβετε την ε, κατάσταση της νησιωτικότητας ως προϋπόθεση για να είναι κανείς επιλέξιμος για τέτοιες κρατικές βοήθειες ε, προκειμένου να αποκατασταθεί η ε, ισότητα ως προς τον ανταγωνισμό των νησιών με άλλες περιοχές και σε ό,τι αφορά την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών προϊόντων σε σχέση με, τα, με τις χώρες που Δυστυχώ, πολύ συχνά παράγουν χωρί να σέβονται τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωση που επιβαρύνουν του ίδιου του Ευρωπαίου παραγωγού. Και τελικά φέρνουν στην αγορά μα προϊόντα με μικρότερο κόστο που φτάνουν στην αγορά μα και είναι πολύ δύσκολο ε, να ανταγωνιστούν οι δικές μας επιχειρήσεις. Μπορούμε να βάλουμε λοιπόν ένα φίλτρο εισόδου είτε με την πρόβλεψη δασμών ή με άλλα μέτρα που θα προστατεύσουν την εσωτερική αγορά και την ανταγωνιστικότητα των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων σε σχέση με τις έξω ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. πολλοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για το θέμα αυτό. Διότι υπάρχει θέμα διαβίωσης, μεταφορικό. Προφανώς είναι δυσκολότερα τα πράγματα σε τέτοιες περιοχές της Ευρώπης. Εργάζομαι περισσότερο σε σχέση με τις εξόχως απόκεντρες περιοχές που βρίσκονται κοντά στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Στις περισσότερες ε, περιπτώσεις, τα νησιά. Εκεί φαίνεται και η διαφορά του σε σχέση με τι εξόχω απόκεντρε. Είναι τελείω διαφορετικέ οι ανάγκε του ω προ τι μεταφορέ, τι εισαγωγέ, προκειμένου να παραμείνουν ανταγωνιστικέ. Και το βλέπουμε και σε άλλε περιοχέ. Δεν μου έρχονται τώρα στο νου νησιά τη Ιταλία. Αλλά αν δείτε τι συμβαίνει με τη Μαδέιρα, λόγω χάρη, έχουμε πολλές ε, περιπτώσεις project, τα οποία έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, προκειμένου να υποστηριχθούν εκεί επιχειρήσεις που δημιουργούν θέσεις απασχόλησης εκεί. Θεωρώ λοιπόν ότι καλά κάνετε και το το θέμα, ε, δεδομένης και της καταγωγής σας. Ε, ε, είμαι έτοιμη να το συζητήσω το θέμα αυτό, διότι αν θεωρείτε ότι υπάρχουν ε, στους καρόνες μας ελλείψεις που δεν προβλέπουν και κάτι για τα νησιά, ευχαρίστως να κάνουμε ένα, ένα ανάλογο τεστ καταλληλότητας για τους κανόνες ε, κρατικής βοήθειας. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να σταθμίσουμε το τι συμβαίνει. Σε ό,τι αφορά τα ευρωπαϊκά προϊόντα, εγώ ίδιος καταναλώτρια, χαίρομαι να μπορώ να βλέπω Πού παράγονται αυτά τα οποία θέλω να αγοράσω ή προτίθεμαι να αγοράσω. Θεωρώ πολύ καλό να βλέπει κανείς που είναι ο τόπος παραγωγής και εγώ βρίσκω ως θετική την ευρωπαϊκή καταγωγή. Τότε έχει κανείς πραγματικά μια επιλογή. Τι κάνουμε τώρα όταν συνάπτουμε εμπορικές συμφωνίες τους δασμούς και αυτό το είδος τους φραγμούς κοιτάζουμε να τους άρουμε, αλλά κοιτάζουμε και να ευθυγραμμίσουμε το τι συμβαίνει, ώστε να αντικατοπτρίζουμε τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Ένωσης. Να υπάρχει δηλαδή δίκαιος ανταγωνισμό, εφόσον κανείς μπορεί να ε, ε, πουλάει τα πρότυπα του εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα πρέπει με τους ίδιους κανόνες να πουλάμε και εμεί τα δικά μας Ε, Υπάρχουν μόνο θέματα με χώρε όπου δεν υπάρχουν εμπορικέ συμφωνίε. Δηλαδή ο μηχανισμός για την ε, κατανάλωση άνθρακα στην παραγωγή ε, είναι κάτι ανάλογο. Ζητάμε από τις ευρωπαϊκές εταιρείες, αυτές που παράγουν στην Ευρώπη, να εξοικονομήσουν ενέργεια, να περιορίσουν την ε, κατανάλωση άνθρακα στην περίπτωση τη παραγωγή του. Δεν μπορούμε να δεχόμαστε εταιρείε εντό Ευρωπαϊκή Ένωση ε, που δεν κάνουν κάτι ανάλογο, εκτό και αν πληρώσουν κάποια αποζημίωση ή για αντιστάθμιση. Τότε υπάρχουν οι κανόνε παιχνιδιού. Δεν έχουν ε, ολοκληρωθεί βεβαίω οι σχετικέ ε, προσπάθειε. Είναι μια συζήτηση που θα γίνει και στο εγγύ μέλλον. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστούμε και την κυρία Αντιπρόεδρο και σας συγχαίρω και για τη δουλειά που έχετε κάνει μέχρι τώρα. Σε όλες τις προηγούμενες παρεμβάσεις ε, υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία ότι η εσωτερική αγορά θα βγει από την κρίση πολύ πιο κατακαιρματισμένη από ό,τι ξεκίνησε. Δηλαδή ότι οι διαφορές ε, μεταξύ ε, κρατών μελών θα είναι μεγαλύτερες στο τέλος της κρίσης από ό,τι στην αρχή. Και υπάρχουν κάποια γεγονότα που κατά την άποψή μου επιβεβαιώνουν ή καταδεικνύουν ότι όντως σωστά ε, ανησυχούμε. Η αρχικά εκεί ω αντίκτυπο της κρίσης δεν ήταν ίδιο για όλε τι χώρε. Κτύπησε κάποιε χώρε πολύ περισσότερο από άλλε. Επίση, οι εθνικέ ενισχύσει συζητήθηκαν πολύ εδώ και εξαρτώνται κυρίω από την ικανότητα και τη διάθεση πόρων που δεν είναι ίδια για κάθε χώρα. Η Γερμανία απορροφά, αν δεν κάνω λάθος, το 51% των ε, ε, ενισχύσεων που εγκρίθηκαν μέχρι τώρα, ενώ υπάρχουν χώρες οι οποίε βρίσκονται το πολύ στο 1% της ε, κρατικής ενίσχυσης. Το πακέτο επίκουσας ανάγκης είναι κυρίως υπομορφή δανείων. Ε, δυστυχώς κάνει παράσιτα ο μιλητής και δεν μπορούμε να ακούσουμε τι λέει. Επίσης, θα πρέπει στο μέλλον να εξασφαλίσουμε και μια κάποια αυτονομία όσον αφορά κάποια προϊόντα ή κάποιους ε, τομείς ενέργειας. Ε, υπάρχει, για παράδειγμα, η πολύ γνωστή περίπτωση της παρακεταμόλης στην Ινδία. Τι γίνεται με την πολιτική ανταγωνισμού και πώς θα μπορέσει να βοηθήσει να υπάρξει αυτή η μεγαλύτερη αυτονομία και η μεγαλύτερη ανεξαρτησία επιμένως σε στρατηγικούς τομείς ε, ε, ο προ... κάτοχός σας, ο κ. Μοσκοβισή, είχε κάποιες ε, ιδέες επ' αυτού και θα ήθελα να ξέρω ποια είναι η δική σας η άποψη. Και τρίτον, στο πρόγραμμα διάσωσης, ανάκτησης, το Recovery Plan, υπάρχουν και κάποια θέματα περιδανείου και να μην σας πω ότι εγώ είμαι υπέρ των μεταφορών και όχι των δανείων ε, και υπάρχουν όροι και ποιοι όροι θα είναι αυτοί σε αυτή την περίπτωση και εγώ να πω ότι προφανώς πρέπει να προσέχουμε ιδιαίτερα όταν χρησιμοποιούμε τα χρήματα όλων. Δυστυχώς ε, κάτι συνέβη με τον ήχο και η δεύτερη σε ε, ερώτηση δεν ε, μεταφράστηκε. Θα απαντήσω λοιπόν στις δύο ερωτήσεις που άκουσα. Πρώτον, όσον αφορά το κατά πόσον θα είναι πιο κατακαιρματισμένη η ενιαία αγορά. Θεωρώ ότι αυτό είναι κάτι το οποίο ανησυχεί πάρα πολλού, ε, και εγώ φυσικά ανησυχώ ε, και γι' αυτό ακριβώς ε, και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα ευρωπαϊκό σχέδιο ανάκτησης και αρχιτεκτονική δομή, αρχιτεκτονική ευρωπαϊκή, γιατί έτσι θα μπορέσουμε να εργαστούμε υπό μια ευρωπαϊκή προοπτική. Και δεύτερον, ήδη πριν από την κρίση είχαμε προτείνει να ξεκινήσει μια task force για την ενιαία αγορά, για να κάνει εκθέσεις για τους φραγμούς της ενέας αγοράς, τι δεν επιτρέπει την βέλτιστη λειτουργία και αυτή η Task Force θα ήταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη ε, για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν αυτούς τους φραγμούς έναν προς έναν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο θα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο και τώρα φυσικά ε, ενώ προετοιμαζόμαστε για να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν οικονομικές ε, ε, ευκολίες για τις επιχειρήσεις, αλλά θα προσπαθήσουμε να μειώσουμε και αυτούς τους φραγμούς, κάποιοι από τους οποίους μπορεί και να αυξήθηκαν λόγω της κρίσης, ακριβώς επειδή ήταν κλειστά τα σύνορά μας. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, διότι η αγορά είναι ένα από τα πιο σημαντικά στοιχεία που διαθέτουμε ε, για την ταχεία και ισχυρή ανάκαμψη, διότι ε, εμπορευόμαστε μεταξύ μας. Ε, έτσι υπάρχει η ανάπτυξη. Ένας επιχειρηματίας μπορεί να έχει προμηθευτές σε μία χώρα και ε, πελάτες σε τρίτη χώρα. Έτσι υποστηρίζουμε τις οικονομίες μας. Η τελευταία ερώτηση όσον αφορά τις εξαρτήσεις Νομίζω εδώ θα πρέπει να δούμε τις σωστές αποχρώσεις, διότι θα ήμασταν πιο φτωχοί και όχι απαραίτητα σε καλύτερη κατάσταση αν ζητήσουμε από όλε τι ε, επιχειρήσεις να εργάζονται μόνο στην Ευρώπη. Αυτό που έχει σημασία είναι ότι σε κάποιους κλάδους υπάρχει μια ε, εξαρτημενωμένη εξάρτηση. Ο συνάδελφος ε, Μπρετών έλεγε ότι πριν από την κρίση υπήρχαν μόνο 10 επιχειρήσεις που παρήγαγαν μάσκες στην Ευρώπη, αλλά τώρα και αυτό φυσικά είναι και προ όφελο του ότι έκανε ο κύριος Μπρετόν, χάρη στα όσα έκανε ο κύριος Μπρετόν, 100 επιχειρήσεις παράγουν μάσκες διότι έγινε μια τεράστια προσπάθεια ώστε να αλλάξει η παραγωγή κάποιων επιχειρήσεων. Και εδώ νομίζω ότι αυτό το οποίο συζητούμε εμεί εσωτερικώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι πώ μπορούμε να έχουμε την απαραίτητη ανθεκτικότητα. Ε, διότι σε αυτού του κρίσιμου τομεί, του οποίου γνωρίζουμε ότι ε, ή θα μπορούσαμε ίσως να συσσωρεύσουμε κάποια πράγματα σε παρκή ε, βαθμό και όταν θα χρησιμοποιηθούν τα αποθέματα να έχουμε χρόνο για να ανακάμψει η παραγωγή ώστε να υπάρξει άλλη πανδημία, αν υπάρξει άλλη πανδημία σαν αυτή που βιώσαμε να είμαστε πιο έτοιμοι. Νομίζω αυτό που έχει σημασία σε επόμενες εβδομάδες είναι να γίνει αυτή η ισορροπημένη συζήτηση, στην οποία θα συζητήσουμε και τι διάφορε αποχρώσει, να πούμε ναι, υπάρχει αυτό ο κλάδο στον οποίο είμαστε πιο ανθεκτικοί και πιο αυτάρκη, αλλά εμεί θέλουμε να είμαστε η Υπήρειο ή η Ένωση, ε, που θα ε, καθορίζουμε του όρου ε, στο εμπόριο. Θέλουμε να είμαστε μια ανοιχτή Υπήρο, διότι πάρα πολλέ επιχειρήσει, πάρα πολλέ θέσει εργασία εξαρτώνται από αυτό. Και αυτό είναι και ένα από του λόγου γιατί ε, του οποίου η Ευρώπη είναι παγκόσμιο παράγων. Ευχαριστώ πολύ. Πόρτα από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Mr. Tang, we cannot hear you. Κύριε Τάγκ, δεν σας ακούμε, λέει ο εκπρόσωπος της γραμματείας. Hello. We can hear you now. Thank you. Ωραία, σας ακούμε τώρα. Προχωρήστε παρακαλώ. Ναι, αλλά δεν ακούει τίποτα ο κύριος Τάγκ. We hear you, Mr. Tank. You can speak. Ο εκπρόσωπος της γραμματείας δίνει το πράσινο φως στον κύριο Τάγκ. Με ακούτε? Ναι, αλλά ο κύριος Τάγκ μάλλον δεν ακούει. Oh, great. <laughs> Sorry for that. Α, ωραία. Εντάξει, αποκαταστάθηκε ο ήχος. Σας ευχαριστώ όλους για τη σημερινή συζήτηση. Εκτιμώ όλη τη δουλειά σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς. Αν και πρέπει να πω ότι η συζήτηση που γίνεται σήμερα στο Ευρωκοινοβούλιο με αφήνει μου αφήνει μια γεύση αμηχανίας. Υπάρχει αθέμητος ανταγωνισμός, άνιση όρη ανταγωνισμού και δεν διαφαίνεται πώς θα μπορέσουμε να υπερβούμε και πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Διότι οι άνισες κρατικές ενισχύσεις που δίνονται αυτή τη στιγμή θα έχουν μακροχρόνιες επιπτώσεις όσον αφορά τη δημιουργία άνισων όρων ανταγωνισμού. Επίσης δεν υπάρχει δίκαιη αποζημίωση, δεν υπάρχουν ε, και προϋποθέσεις αν θέλετε για την παροχή κρατικών ενισχύσεων, βραχυπρόθεσμες ίσως αλλά όχι μακροπρόθεσμες. Άρα πιθανότητα εμείς ως πολίτες, ως φορολογούμενοι θα επομιστούμε το κόστος αυτών των κρατικών ενισχύσεων χωρίς να υπάρχει κάποιο όφελος. Υπάρχει κάποιος κανόνας, υπάρχει κάποια πρόβλεψη αποζημίωσης στους κανόνες αυτούς. Δεν θα μπορούσαμε για παράδειγμα να ζητήσουμε από τις εταιρείε που έχουν λάβει κρατικές ενισχύσεις να καταρτήσουν ένα σχέδιο μετάβασης για το πώς δηλαδή θα ε, επιστρέψουν αν θέλετε τα χρήματα που έχουν λάβει με τη μορφή κρατικών ενισχύσεων από εμάς τους φορολογούμενους πώς θα τα επιστρέψουν με τρόπο που θα αποβαίνει σε όφελος των ίδιων των φορολογουμένων και των πολιτών. Η κυρία Βεστάγκερ. Σας ευχαριστώ. Είναι θετικό το γεγονός ότι επανερχόμαστε σε αυτό το ζήτημα, διότι το να, υπάρχουν, να υπάρχει δικαιοσύνη, να υπάρχουν ίσοι όροι ανταγωνισμού, το να μπορεί κανείς να έχει ευκαιρίες όσον αφορά την παραγωγή, την έρευνα, την καινοτομία για το πώς μπορεί κανείς να, παράγει, να παράσχει τα προϊόντα του στους καταναλωτές. Αυτά όλα είναι τα ουσιώδη, ουσιώδη θέματα. Και στην έκθεση για τον ανταγωνισμό υπάρχει πραγματικά ιδιαίτερα τονισμένη αυτή η διάσταση του δίκαιου, του, του ανταγωνισμού. Εμείς διακρίνουμε μεταξύ ενισχύσεων ρευστότητας που κατευθύνονται σε επιχειρήσεις προκειμένου να μπορέσουν να ε, επιβιώσουν την καραντίνα και αφενός δηλαδή και αφετέρου σε ενισχύσεις που δίνει τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις να έχει τη δυνατότητα όχι ως πρώτο μέτρο αλλά ως έσχατο μέτρο να ζητηθεί βοήθεια δηλαδή προκειμένου να ε, διασφαλιστεί η κεφαλαιακή της επάρκεια. Για όλα αυτά τα θέματα βεβαίως προτού εγκρίνουμε τις συστάσεις και τους κανόνες αυτούς έχουμε διαβολευτεί εκτενώς με τα κράτη-μέλη και αυτά που χρειάστηκε να εξωσορροπήσουμε ήταν ακριβώς αφενός πώς θα εξασφαλίσουμε ότι οι φορολογούμενοι θα ωφεληθούν για τον κίνδυνο, για το ρίσκο που καλύπτουν αυτών των επιχειρήσεων. Διότι γιατί για τις μεγάλες ειδικά επιχειρήσεις οι εγγυήσεις που δίνονται είναι πάρα πάρα πολύ ψηλές. Ταυτόχρονα θέλαμε να δώσουμε κίνητρο στις επιχειρήσεις ώστε τα κρατικά κεφάλαια να αποχωρήσουν όσο το δυνατόν γρηγορότερα για να ορθοποδήσουν και πάλι. Γι' αυτό και ε, έχουμε βάλει κανόνες όσον αφορά τα μπόνους, τα μερίσματα για τους μετόχους, για τις, ε, τα προγράμματα επαναγοράς μετοχών, οπότε όσο το κράτος συμμετέχει με τις ενισχύσεις αυτές, ο πρώτος που θα αποζημιωθεί, που θα υποφεληθεί θα είναι ο φορολογούμενος. Αυτό είναι το πρώτο στοιχείο. Δεύτερο στοιχείο είναι η διαφάνεια. Ξέρετε ότι οι μεγάλες επιχειρήσεις που λαμβάνουν ε, κρατικές ενισχύσεις θα πρέπει να λογοδοτήσουν για το πώς θα αξιοποιήσουν και θα χρησιμοποιήσουν τη βοήθεια αυτή. Τέλος, αν είσαι μεγάλη εταιρεία και πάρεις κρατική ενίσχυση, υπάρχουν, ζητούμε εγγυήσεις για το πώς η πιθανή στρέβλωση της αγοράς και του ανταγωνισμού θα ε, αντισταθμιστεί. Γιατί υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες δεν θα μπορέσουν να πάρουν τέτοιες, τέτοιες ενισχύσεις. Γι' αυτό και στο προσωρινό πλαίσιο έχουμε θεσπίσει κανόνα ότι οι εταιρείε με δεσπόδους θέση στην αγορά θα πρέπει να το λαμβάνουν αυτό υπόψη τους, διότι διαφορετικά δεν θα μπορούν να τις ανταγωνίζονται μικρότερες επιχειρήσεις, άπαξ και ξεπεράσουμε αυτήν την κρίση και επανέλθουμε σε μια κάποια κανονικότητα. Ευχαριστούμε κυρία Στεφανή Ουρτών από τους Η κυρία Γιώκουρτα. Η κυρία Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε. Κυρία Φεστάγκερ, είναι πάντα χαρά μας να βρισκόμαστε ακόμα και από απόσταση. Για το θέμα του οποίου ήμουν εισηγήτρια δεν μπόρεσε να συζητηθεί ούτε να ψηφιστεί λόγω της, ολομέλειας, των ακυρώσεων στην Ολομέλεια του Μαρτίου και της κρίσης του κορονοϊού πάντω να σα ενημερώσουμε ότι θα προσπαθήσουμε να υποβάλουμε νέε τροπολογίε για να ενισχυθεί η έκθεση αυτή και υπό το φω των εξελίξεων ε, τη κρίσης του κορονοϊού. Θα εργαστούμε τι ε, εβδομάδε, ε, τι επόμενε με τους κοιόδης εισηγητέ για να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ευχαριστώ του συναδέλφου για την εξωσημείωτη δουλειά της Επιτροπής τη δική μα και τη δική σα και των συνεργατών σα. Έχετε θίξει δύο ζητήματα. Και θέλω να το σχολιάσω και εγώ. Το είπατε κι εσείς και θα το είπαν κι άλλοι συνάδελφοι, πρόεδρε. Η ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στρατηγικού τομεί τη έχουν πληγεί λόγω του κορονοϊού. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να ξαναβρει την οικονομική τη επικυριαρχία ε, ανασυγκροτώντας τα συγκριτικά τη πλεονεκτήματα σε τομεί κλειδιά. Τομεί όπου είμαστε εξαρτημένοι από τι εισαγωγέ πάρα πολύ σήμερα. Όπω στην ε, φαρμακοβιομηχανία. Η πολιτική ανταγωνισμού είναι ένα καθοριστικό εργαλείο για να βεβαιωθούμε ότι η πολιτική αυτή της οικονομικής επικυριαρχίας, της πολιτικής και βιομηχανική επικυριαρχίας ε, που επιτρέπει τη βολονταριστική προσέγγιση, διασφαλίζεται ακόμα. Ε, σε σχέση λοιπόν με όσα είπε ο συνάδελφό σα για την εσωτερική αγορά, ο κ. Μπρετό, Πώ θα βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα και διαφυλάσσεται αυτό εφόσον έχει στρατηγική σημασία και μετά για τον έλεγχο των ε, συγκεντρώσεων και των συγχωνεύσεων. Ένα σημαντικότερο θέμα θα μπορούμε να επιτρέπουμε συγχωνεύσεις και συγκεντρώσεις ε, σε σχέση με το failing defense για να ε, δούμε πώς πρέπει να προστατευτούν κάποιες εταιρείε στα πλαίσια της κρίσης του κορονοϊού. Θα πρέπει ενδεχομένως οι αυστηρές συνθήκες ε, των συγχωνεύσεων και συγκεντρώσεων να επαναθεωρηθούν εφόσον κάποιες φορές καθιστούν οποιαδήποτε κίνηση πάρα πολύ δύσκολη. Πολλέ εταιρείε πτώχευση θα ζητήσουν ε, τέτοια εξαγορά ή τον επιτραπούν οι συγχωνεύσει τους. Και πάλι στη στο θέμα των συγκεντρώσεων, τι θα γίνει σε σχέση με τις ε, σχετικές αγορές και την αναθεώρηση των κανόνων τους. Πώς έχει προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τι περιμένετε από το Κοινοβούλιο και την Επιτροπή ΕΚΟΝ προ αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ πολύ. Και πάλι ευχαριστούμε για τη δουλειά που κάνατε, για την έκθεση, για τον ανταγωνισμό. Πραγματικά ανυπομονώ για να γίνει συζήτηση και στην Ολομέλεια. Και νομίζω ότι είναι πολύ επίκαιρο να το συζητήσουμε για να, να απηχηθούν όσα συμβαίνουν τώρα και στην μελλοντική έκθεση ανταγωνισμού. Θα γίνει και πιο σημαντική έτσι. Θέλω να δω και τι τροπολογίες θα προτείνετε λοιπόν. Η εξάρτηση που μας απασχολεί έχει να κάνει κυρίως με, κάποιο με τον τομέα των φαρμακοβιομηχανιών βεβαίως. Και όπως είπα αρχικά, το πλαίσιο για τη συνεργασία έχει να κάνει και με την παραγωγή φαρμάκων. Κάποια γενώσιμα είδαμε ότι μπορεί να εξέλιπαν. Όχι αναγκαστικά από τα ακριβότερα ή από τα πιο δυσέβρετα, αλλά επειδή ξαφνικά έγινε τεράστια ζήτησή τους, ήταν σημαντικό για τις εταιρείε να μπορούν να συνεργαστούν για να υπάρξει επαρκής προσφορά. Είναι σημαντικό αυτό. Όταν μιλάμε για κάποια από τα βασικά μόρια, και για την ε, προσφορά επί τις οποίες μπορούμε να βασιστούμε. Προς στιγμήν δεν είχαμε καμία επαφή για το Failing Firm Defense, για την ε, εταιρεία σε πτώχευση που πρέπει να προστατευτεί. Οι κρατικέ βοήθειες που δίδονται τώρα έχουν πετύχει. Μπορεί να υπάρχουν αναχώρα παραδείγματα βεβαίω που δεν γνωρίζω ακριβώ, όπου κάποια όρια που έχουμε θέσει το επίπεδο τη Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχουν χρησιμοποιηθεί σωστά. Δεν ξέρω αυτή τη στιγμή που μπορεί να υπάρχουν ζητήματα που μπορεί να είναι προβληματικά. Θα ξέρετε πάντω ότι στο σχετικό πλαίσιο έχουμε πει ότι μόνο από εξαιρετικέ προποθέσει μπορεί μια εταιρεία που υποστηρίχθηκε στο κεφάλαιό τη να αγοράσει άλλε εταιρείε. Διότι φοβούμεθα ότι αυτό μπορεί να στρεβλώσει τους κανόνες ανταγωνισμού. Τώρα για, την, ε, ε, για τον ορισμό μιας αγοράς θα πρέπει να ξεκινήσουν δημόσιες διαβουλεύσεις. Δεν έχω ακόμη το χρονοδιάγραμμα. Απλώς κοιτάζουμε, όπως ξέρετε, όλους τους κανόνες μας, της κρατική βοήθειας και μια σειρά αποζητήματα. Το τελευταίο που είχα ανακοινώσει είναι ότι θα δούμε και τις κατευθυντήριες γραμμές μας για το διαδικτύου. Κάτι που ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί στι αρχές του καλοκαιριού. Και μετά θα υπάρξουν δημόσιε διαβουλεύσει για κάποια από αυτά τα ζητήματα. Ευχαρίστω να επανέλθω και να σα δώσω ακριβέστερε πληροφορίε για το πρόγραμμα, αλλά η δουλειά αυτή είναι σε εξέλιξη παρά την πίεση που ασκεί η κρίση του κορονοϊού. Ελπίζω λοιπόν ότι θα μπορέσω να επανέλθω σύντομα. Thank you very much. Now we have... Ευχαριστώ πολύ. Τώρα έχουμε κάποια αιτήματα για τη διαδικασία Catch the Eye. Έχουμε 7 λεπτά μόνο στη διάθεσή μας. Επομένως, θα συγκεντρώσουμε λίγο στα γρήγορα όλες τις ερωτήσεις, ένα λεπτό για τον καθένα και μετά θα δώσει μια σύντομη απάντηση η Αντιπρόεδρος Βεστάγκερ. Ο Σβεν Γίγκολ πρώτα. Ευχαριστώ Κυρία Πρόεδρε, ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Κρίμα που δεν μπορούμε να σας δούμε διαζώσεις. Έχω δύο πολύ συγκεκριμένε ερωτήσεις. Πρώτον, έγινε πολύ ντόρος ε, για την κατανομή της συγκεκριμένη κρατικής ενίσχυσης από τα κράτη-μέλη. Μπορείτε να μας ενημερώσετε για τα μερίδια του κάθε κράτους μέλους με τα πιο πρόσφατα στοιχεία. Και επίση, θα μπορούσατε να δεσμευτείτε να δημοσιεύετε εβδομαδιαίες επικαιροποίησεις ε, της κρατικής ενίσχυσης που εκκρίθηκε από κάθε κράτος μέλος. Θα το εκτιμούσαμε ιδιαίτερως για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε και τη δημόσια συζήτηση για τα μέτρα στην κοινή αγορά. Και δεύτερον, μία απλή ε, ερώτηση. Δεν θα ήταν πιο σωστό να ζητούμε από τις επιχειρήσεις που λαμβάνουν κρατική ενίσχυση να δημοσιεύουν αναχώρα που κατέβαλαν ε, φόρους που ε, ε, έκαναν έσοδα και που τα κατέγραψαν. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ Σβέν. Ο Λευτέρης Νικολάου Αλαβάνος τώρα από τους μη We cannot hear you. Um... Δεν σας ακούμε. Μπορείτε να κάνετε ένα refresh στη σελίδα. Can you hear me now? Now we can hear you, thank you. Ακούτε τώρα. Λοιπόν, στο σύντομο χρόνο που έχω στη διάθεσή μου θα ήθελα να αναφέρω δύο πτυχές μια πολύ σύνθετη κατάσταση. Καταρχάς, όσον αφορά την πανδημία του COVID-19 υπάρχει μια πτυχή που αφορά την ε, υγειονομική κρίση ε, σε τι συμπέρισμα καταλήγουμε όσον αφορά ε, την κατάσταση στην Ευρώπη και παγκοσμίω. Αυτό που χρειαζόμαστε είναι πραγματικά εύρωστα κρατικά συστήματα που εγγυώνται ε, το δικαίωμα όλων των πολιτών σε κάθε χώρα σε υγειονομική περίθαλψη. Πώς έχει κατάσταση τώρα μετά από την σταδιακή άρση των διαδικασιών των μέτρων ε, είναι η κατάσταση χειρότερη ή καλύτερη από πριν. Και τι έγινε με τις ενισχύσεις οι οποίες δόθηκαν για να είναι πιο ανθεκτικό το κρατικό σύστημα υγείας. Τίποτα, γιατί τα περισσότερα πήγαιναν σε ε, ενισχύσεις ιδιωτικών δομών υγείας. Το δεύτερο έχει ε, σχέση με την κατάσταση των εργαζομένων και το τι αντιμετωπίζουν. Έχουμε απολύσεις, έχουμε αρνητικές ε, ε, εξελίξεις σε συλλογικές συμβάσεις και αυτή η κατάσταση δεν θα βελτιωθεί με όλες αυτές τις ε, προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, και της Ευρωπαϊκής Ένωσης εν γέννη. Ε, υπάρχουν με προγράμματα τα οποία δεν βοηθούν στην ουσία τους εργαζομένους. Δείτε τι γίνεται στην Ελλάδα. Εν μέσω της πανδημίας του COVID-19 έχουμε την κυβέρνηση να, προκύπτει, να προτείνει περαιτέρω περικοπή των μισθών μέχρι και 10%. Ο κόσμος πλήρωσε το τίμημα για την προηγούμενη κρίση και τώρα θα υποχρεωθούν να πληρώσουν και μια, ένα επόμενο τίμηνο. Δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο. Ευχαριστώ. Να τηρείτε το χρόνο του ένα λεπτό. Ο Πιέρ Νικόλα Πεντιτσίνη τώρα, πάλι μία εγγεγραμμένο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε Βεστάγκερ, η ότι μέχρι τώρα έχετε εγκρίνει 175 μέτρα κρατική ενίσχυση συνολική αξία 2-3 ευρώ. Αλλά ξεχάσατε να υπενθυμίσετε ότι το 51% ε, είναι για τη Γερμανία. Λοιπόν, ε, μέσω μιας συμμετρικής κρίσης εγκρίθηκαν ασύμετρα μέτρα τα οποία θα υποχρεώσουν ε, για άλλη μια φορά χώρες που δεν έχουν φορολογικό ε, περιθώριο ε, να βρεθούν σε μειονεκτική θέση σε σχέση με τις άλλες χώρες. Και πάλι κερδισμένη είναι η Γερμανία. Ένα τρεις για μία χώρα και άλλα ένα τρεις για μία υπόλοιπη ήπειρο. Ε, η Γερμανία ήδη παραβιάζει τους κανόνες ε, για το πλεόνασμα χωρίς καμία διαδικασία επιπαραβάση και κανένα δικαστήριο δεν κάνει κάτι για την παραβίαση της αρχής αναλογικότητας. Κυρία Επίτροπε, λοιπόν, δεν έχουμε τίποτα το καινούριο εδώ. Αν δεν μπορέσετε να εφαρμόσετε διορθωτικά μέτρα για αυτές τις αδικίες, ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα είναι συνυπεύθυνη για την κατάσταση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάρκες από το S&D. Ε, Ευχαριστώ. Με ακούτε? Ναι, σας ακούμε, αλλά δυστυχώς δεν σας βλέπουμε. Να προσπαθήσω. Με βλέπετε? Όχι. So Υπάρχει πρόβλημα με το βίντεο, αλλά μπορώ να μιλήσω μάλλον. Σωστά. Ωραία. Η πρώτη με ερώτηση προς την κυρία Βεστάγκερ, την Αντιπρόεδρο, ε, είναι ότι πρώτον, αυτό σας ευχαριστήσω για την παρουσίασή σας, να πω ότι μιλήσατε για φόρο στα ψηφιακά έγινε μια τέτοια συζήτηση. Συμφωνείτε ότι οι φόροι για τα ψηφιακά θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να χρηματοδοτηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πώς. Με ενδιαφέρει ιδίω η απάντησή σας για το θέμα αυτό, ε, καθώς είμαι συνεισηγήτρια για το θέμα του πολιτιούς δημοσιονομικού πλαισίου. Και έπειτα, ως πότε η ευελιξία στις κρατικές βοήθειες θα ισχύει, διότι Τάλθηκαν οι κανόνε για τι κρατικέ βοήθειε. Μπράβο σα, Επιτροπή, που μέχρι τώρα δεν εφαρμόζονται του ίδιου αυστηρού κανόνε. Όμω, όπω και άλλοι συνάδελφοι το είπαν προηγουμένω, με ενδιαφέρει κατά πόσον οι αποκλήσει που δημιουργήθηκαν μεταξύ 100 μελών θα καλυφθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτηκε στα πλαίσια του προγράμματο ανάκαμψη να κοιτάξει και μια πολιτική παράμετρο για να ξαναυπάρξουν ίσοι κανόνες ανταγωνισμού στην εσωτερική αγορά. Το ερώτημα είναι τι στρατηγικές θα προκρίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τι θα επιδιώξει ώστε να βεβαιωθεί ότι το πρόγραμμα αυτό πραγματικά θα οδηγήσει στην σύγκληση και να υπάρξει το λεγόμενο level playing field, δηλαδή σε κανόνες παιχνιδιού και όχι αυτές οι αποκλήσεις που παρατηρούμε τώρα μεταξύ των κρατών μελών. Ευχαριστώ. Now we have Fabio Massimo Castaldo, please. Και τώρα... Έχουμε τον... Και τώρα ο κύριος Καστάλντο, διότι αν δεν βλέπετε, ε, αν δεν σας βλέπουν οι μεταφραστές δεν μπορείτε να μεταφράσετε. Φάμπιο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστώ Ιρένε, ευχαριστώ την Αντιπρόεδρο Βεστάγκερ για τις παρατηρήσεις που μα έκανε σήμερα. Είμαι πεπισμένο ότι αυτή η οικονομική κρίση του κορονοϊού 2019 δεν θα είναι μόνο ένα μακροοικονομικό πρόβλημα, ίσω και μια ευκαιρία για να καλύψουμε κάποιε ασυμμετρίε που υπάρχουν τώρα στο εσωτερικό τη εσωτερική αγορά. Ιδίω για κάποιου που εκμεταλλεύονται τα πλεονεκτήματά του χωρί να πληρώνουν τίποτα. Άκουσα το γεγονό ότι εσεί θα είσαστε υπέρ ενό φόρου στα ψηφιακά, ενό από του τομεί που δεν έχουν πληγεί από την κρίση και μάλιστα έχουν ευνοηθεί. Οι μεγάλε εταιρείε, οι γιγαντιέ εταιρείε του ψηφιακού τομέα έχουν ευνοηθεί. Ε, και λόγω των φορολογικών κανόνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, πληρώνουν τον ελάχιστο από το φόρο που οφείλουν. Ε, εδώ όμω αυτό με φέρνει και σε ένα άλλο θέμα. Το θέμα των επιθετικών φορολογικών συμφωνιών που έχουν ε, διοργανώσει κάποια κάποια μέλη, ε, καταλυστεύοντα όμω έτσι του πόρου άλλων κρατομελών. Δηλαδή, εδώ μιλάμε για συνενοχή σε ένα συλλογικό ε, παιχνίδι που ουσιαστικά αποσπά τα κέρδη των φορολογουμένων φορολογική παράδειση, με συμφωνίες όπως η CCCTB, η CBCR, πράγματα που αποδυναμώνουν την ενιαία αγορά. Δεν είναι κάτι που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Με την πρόταση που θα μα κάνει η κυρία Φόντερ Λάιν την Τετάρτη, δεν πρέπει κάτι να περιμένουμε σχετικά. Ελπίζω τώρα να υπάρξει η θέληση να προχωρήσουμε σωστά για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα έλλειψη ε, ε, ισότητα και εσύ αντιμετώπιση από τη δικαιοσύνη στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει ε, και τα κράτη, τα κράτη να μπορέσουν να ωφεληθούν αναλόγω από του κανόνε που βλέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα που δεν αφορά άμεσα τις αρμοδιότητες σας, όμως επειδή η πανδημία αυτή έχει πλήξει την ενιαία αγορά, θέλω να ρωτήσω αν η Κομισιόν έχει πληροφορίες σχετικά με την πηγή, την προέλευση αυτού του ιού. Και πιο συγκεκριμένα, γνωρίζετε τι συμβαίνει σχετικά με έρευνες για παθογόνους ιούς. Έχετε συζητήσει ε, αυτό το θέμα. Θα το διερευνήσετε αυτό το θέμα. Διότι υπάρχουν ε, πειράματα τα οποία ε, γίνονται για, σε παθογόνους μικροοργανισμούς και δεν αποκλείεται ενδεχομένως και αυτή η πανδημία με τις τόσο σοβαρές επιπτώσεις της να έχει προέλθει από κάποιο τέτοιο εργαστήριο. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αιναλουόμα. Καλησπέρα και σας ευχαριστούμε κυρία Βεστάγκερ για την πολύ σημαντική και απαιτητική δουλειά που κάνετε και πρέπει να πω ότι εσείς και το επιτελείο σας έχετε φανεί εξαιρετικά αποτελεσματικοί. Αξιοθαύμαστο. Πρώτον, έχω δύο ερωτήσεις. Πρώτον, Ταμείο Ανάκαμψης Κρατικών Ενσχύσεων. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει ένα τέτοιο ταμείο. Όμως αυτό που θα με ενδιέφερε να μάθω είναι αν κονδύλια από αυτό το Ταμείο Ανάκαμψης θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως κρατικές ενισχύσεις για τις επιχειρήσεις. Και δεύτερο ερώτημα είναι το εξής. Όταν υπάρχει υπερπροσφορά σε κάποιον κλάδο, όπως για παράδειγμα στον κλάδο των αερομεταφορών, πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα δοθούν κρατικές ενισχύσεις σε διάφορες εταιρείες ώστε ακριβώς να μην συνεχιστεί μια κατάσταση υπερπροσφοράς. Γιατί νομίζω ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν ιδιαίτερα σόφρον όσον αφορά την αξιοποίηση των ε, χρημάτων των φορολογουμένων. Πρόεδρος, ευχαριστώ. Fitzgerald, τελευταίος ομιλητής. Τελευταίο ομιλήτρια. Hello, you can hear me. Γεια σας, με ακούτε. Ναι, σας ακούμε, λέει η γραμματεία. Ευχαριστούμε, Επίτροπε, εσάς και το επιτελείο σας για όλη τη δουλειά που έχετε κάνει. Θέλω να θέσω ένα ερώτημα σχετικά με τις, αερομετα με τις αεροπορικές εταιρείες. Κάποιες από αυτές έχουν ε, λάβει κρατικές ενισχύσεις, ε, πακέτα διάσωσης. Και θέλω να ρωτήσω τα εξής σε σχέση με αυτό το θέμα. όταν θα ξαναξεκινήσουν οι πτήσεις, θα μπορούσαν ενδεχομένω κάποιες ε, εταιρείε, χάρη στις κρατικές ενισχύσεις που, που δόθηκαν, να προσφέρουν τα εισιτήριά τους σε πολύ χαμηλή τιμή. Αυτό δεν θα είναι στρέβλωση του ανταγωνισμού. Πώς η Κομισιόν θα εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρξει περαιτέρω στρέβλωση, αν θέλετε. Δεύτερο ερώτημα. Όταν επανέλθουν οι αεροπορικές εταιρείε στην κανονικότητα, πώς θα εξασφαλίσετε ότι οι κρατικές ενισχύσεις που δόθηκαν στις εταιρείε αυτές πράγματι αφορούσαν μόνο τη διάρκεια της πανδημίας, δεδομένης και της χαλάρωσης των ε, κανόνων κρατικών ενισχύσεων. Φαντάζομαι ότι θα, θα έχετε κάποιους μηχανισμούς ήδη, απλά θέλω να μου το ε, επιβεβαιώσετε. Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ. Αυτά όσον αφορά τη διαδικασία Catch the και τις ερωτήσεις. Ζητώ συγγνώμη από την Αντιπρόεδρο αν τελικά χρειαστήκαμε ε, λίγο παραπάνω. Διερμηνία θα έχουμε για άλλα 9 λεπτά αν θέλετε κυρία Βεστάγερ, έχουμε λίγη ώρα ακόμη για να μας δώσετε τις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τους διερμηνείς. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι εξαιρετικό το γεγονός ότι έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Ιδάλλως πραγματικά θα ήμουν χαμένη, διότι οι γλωσσικές μου δεξιότητες φυσικά δεν αρκούν για να παρακολουθώ τους πάντες. Όσον αφορά την ερώτηση του Σφέν έχουμε 177 εθνικά μέτρα αυτή τη στιγμή που αναλογούν σε 2,3 τρισεκατομμύρια ευρώ περίπου. Αυτό φυσικά συνοδεύεται και από πολύ σημαντικές δικλείδες ασφαλείας, διότι αυτός είναι ο προπολογισμό αυτών των προγραμμάτων και δεν ε, έχουν συγκεκριμένο προϋπολογισμό όλα τα προγράμματα και δεν είναι δεδομένο ότι θα καταβληθεί όλο ε, ο προπολογισμό. Πρέπει λοιπόν να τα θεωρούμε ως ε, συνολικά ποσά, όχι ακριβώς τα ποσά τα οποία καταβλήθηκαν ή καταβάλλονται. Από αυτά τα 2,3 τρισεκατομμύρια που έχουμε ως εκτίμηση, το 47% το έχει πάρει η Γερμανία, η Ιταλία περίπου 18%, η Γαλλία 16%, η Ισπανία πάνω από 4%, το Ηνωμένο Βασίλειο περίπου 4%, η Πολωνία περίπου 2,5%, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη είναι 1,5% ή και χαμηλότερα. Δεν θεωρώ ότι η εβδομαδιαία επικαιροποίηση θα αλλάζει πάρα πολύ αυτά τα στοιχεία, αλλά βεβαίως πολύ ευχαρίστως ε, να επανέλθω, διότι όπως σας είπα, η διαφάνεια για το πού πηγαίνουν αυτά τα κονδύλια είναι ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία για μας. Γι' αυτό και ακριβώς ζητούμε διαφάνεια και σε μεμονωμένες αποφάσεις, ώστε οι πολίτες και ο τύπος, οι δημοσιογράφοι στα κράτη-μέλη να μπορούν να παρακολουθήσουν τι συμβαίνει. Κάποια κράτη-μέλη ζητούν από τις επιχειρήσεις απλώς να υποβάλουν ε, στοιχεία για ενίσχυση μόνο αν καταβάλουν φορολογία στο κράτος μέλος. Αυτό ε, δεν νομίζω ότι μπορούμε να το κάνουμε εμείς ε, λόγω της νομικής βάσης που έχει καθοριστεί αρχικώς όσον αφορά το θέμα αυτό. Αλλά πέραν αυτού υπήρξαν και κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά την ψηφιακή φορολόγηση. Ανεξάρτητα από το τι θα συμβεί ε, με τα έσοδα από ένα ψηφιακό φόρο, θεωρώ ότι είναι υψής της σημασίας κάθε επιχείρηση να καταβάλει ένα τέτοιο φόρο. Ε, τώρα διαπιστώνουμε ότι πολλές από τις επιχειρήσεις που καταβάλουν ε, τους φόρους τους σε μεγάλο βαθμό συνέβαλαν και σε αυτές τις κρατικές ενισχύσεις που δίνονται. Ε, και είναι πάρα πολύ σημαντικό οι επιχειρήσεις οι οποίες διεξάγουν τις δραστηριότητες τους στην Ευρώπη να βοηθήσουν και στην ανάκαμψη από όλα τα κράτη-μέλη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Εγώ προσωπικά εκτιμώ και τους ίδιους πόρους ε, όσον αφορά την ψηφιακή φορολόγηση, αλλά για μένα αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να υπάρξει για ε, ε, τη διαχείριση της φορολογίας και για τις πάρα πολλές επιχειρήσεις που ούτως ή άλλως ήδη καταβάλουν τους φόρους τους. για την ερώτηση του κυρίου Νικολάου Λαβάνου. σε αυτούς τους πολύ δύσκολους καιρούς ε, εκτίμησα το ιδιαίτερο στο γεγονός ότι ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει καθολική πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Νομίζω ότι ένα από αυτά τα οποία έχουμε καταφέρει με τις προσπάθειες, τις τεράστιες προσπάθειες των πολιτών σε κάθε κρατος μέλος, αυτούς που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, γιατρούς, ε, νοσοκόμους, υγειονομικό προσωπικό και κόσμο στις μεταφορές και στο λιανεμπόριο, είναι ότι όχι μόνο σώθηκαν ζωές, αλλά σώθηκε και το κοινωνικό συμβόλαιο, ότι υπάρχει ένα σύστημα υγείας για σας εάν αρρωστήσετε, ότι το σύστημα υγείας δεν καταραίει, δεν ε, ε, υποβαθμίζεται, αλλά υπάρχει ένα σύστημα υγείας. Και νομίζω ότι με αυτές τις τεράστιες προσπάθειες τα καταφέραμε. Όσον αφορά το γεγονός ότι ε, τα προγράμματα στήριξης ε, ε, για την ανεργία μόλις τώρα εγκρίθηκαν και τώρα αρχίζουν να εφαρμόζονται, από 1η Ιουνίου δηλαδή θα εφαρμοστεί, γι' αυτό ίσως δεν έχει δει οι εργαζόμενοι κάποια αποτελέσματα. Βέβαια είναι ένα θέμα το οποίο ανακύκτει συνεχώς και πραγματικά ε, σας συγχαίρω που ε, επιμένετε σε αυτό το σημείο το, να, ε, το γεγονός ότι είναι, δεν είναι ισότιμη η ώρα ανταγωνισμού. Δείτε τα πράγματα από μια άλλη προοπτική. Εδώ και χρόνια ζητούσαμε τη Γερμανία να δαπανά περισσότερο τώρα δαπανούν περισσότερο και νομίζω ότι εμέσως αυτό ε, βοηθά και κάποιες άλλες επιχειρήσεις εκτός Γερμανίας. Γιατί οι γερμανικές επιχειρήσεις είναι τμήμα της ε, αλυσίδας ε, διανομής της Ευρώπης. Ε, έχουν προμηθευτές, πελάτες σε σχεδόν όλες τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Και φυσικά αυτό είναι στοιχείο της εξίσωσης. Δεν αναιρεί το γεγονός ότι θα μπορούσε να υπάρχει και κίνδυνος κατακαιρματισμού της αγοράς, αλλά είναι τμήμα της εξίσωσης. Το να δαπανά τόσο πολλά ένα μεγάλο κράτο μέλη είναι και κάτι το οποίο δίνει τη δυνατότητα για την αλυσίδα διανομή ε, την οποία ε, χρειάζονται οι επιχειρήσει και στην οποία συμμετέχουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης, όπως γνωρίζετε, έχει ξεκινήσει και την ε, ρήτρα διαφυγής που δίνει τη δυνατότητα για μεγαλύτερα περιθώριο δανεισμού στον εθνικό προπολογισμό. Και τέλος, κατ' εξίσου σημαντικό, αν δείτε το προσωρινό πλαίσιο, δεν μπορούμε να εγκρίνουμε ενίσχυση η οποία δεν θα είναι αναλογική. Επομένως, ακόμα και σε χώρες όπου ε, δίνεται πολλή ενίσχυση, είναι αναλογική. Δεν είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνει γίνεται ε, σε μια ε, οξία κρίση. Και αυτό σημαίνει ότι ακόμα και όταν πρόκειται για ανακεφαλαιοποίηση, αυτή θα είναι ανακεφαλαιοποίηση για την ε, αποκατάσταση του κεφαλαίου της προηγούμενης χρονιάς. Δεν είναι κάτι το οποίο θα δώσει τη δυνατότητα σε κάποιον να κάνει κάτι το οποίο δεν θα είχε κάνει σε άλλη περίπτωση. Και νομίζω ότι το γεγονός ότι υπάρχουν και κάποια όρια ε, έχουμε, μας επιτρέπει να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση που θα μειώσει τη στρέβλωση του ανταγωνισμού ε, και δεν θα μπορεί να κάνει κάποιος ε, εξαγορά ξέρω επιχειρήσεων με μερίσματα. Υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι φυσικά και για τους μετόχους ώστε οι πιθανές στρεβλώσεις ανταγωνισμού από επιχειρήσεις οι οποίες θα ήθελαν να κάνουν κάτι τέτοιο να προστατεύουν τις υπόλοιπε. Ελπίζω ότι το σχέδιο το οποίο θα παρουσιάσουμε την Τετάρτη θα είναι και τμήμα της απάντησης. Πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να υπάρξει μια ευρωπαϊκή ανάκαμψη, να είναι ισχυρή αυτή η ανάκαμψη και να έρθει γρήγορα. Και πραγματικά ελπίζω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα κάνει αυτό που κάνει πάντα. Δηλαδή να επικεντρωθεί σε αυτό και να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει αυτό πολύ γρήγορα ε, στις διαπραγματεύσεις. Βεβαίως ε, θα πρέπει να αποτελέσει και πηγή έμπνευση για, για τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων ε, ελπίζω να μπορέσουν σύντομα να συναντηθούν και διαζώσεις για να μπορέσουν να κάνουν τις διαπραγματεύσεις. Όσον αφορά την εμπειρία, στην πορεία του ιού, δεν έχω ακούσει τίποτα το οποίο να υποστηρίζει μια τέτοια ιδέα. Ε, απολύτως τίποτα. για τις αεροπορικές εταιρείε ε, και ε, τις υπερβολικές ε, δυνατότητες, αυτό δεν είναι υποσυζήτηση αυτή τη στιγμή. Αν είναι επιχειρήσεις οι οποίες είχαν δυσκολίες πριν από την 1η Ιανουαρίου, μπορούν να λάβουν αποζημίωση για ζημίες, αλλά δεν μπορούν να λάβουν κρατική ενίσχυση αυτή καθεαυτή. Και φυσικά η αγορά ε, θα το γνωρίζει και με τις αβεβαιότητες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ δύσκολο να προβλέψει ε, ποιο θα είναι το μέλλον ε, των αεροπορικών μεταφορών. Μπορεί να ε, επιδοτείται για αρκετό καιρό, ακόμα και αν ανοίξουν ε, σιγά σιγά τα και όταν θα ανοίξουν σιγά σιγά τα σύνορα. Τέλος, ε, Ξέρετε ότι εκτιμώ ιδιαίτερα τη συνεργασία μαζί σας και προσβλέπω φυσικά σε μια εσβάθος συζήτηση όταν ε, θα ε, παρουσιαστεί η δέσμη μέτρων την Δετάρτη. Αλλά αυτό το οποίο ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μένα είναι ότι χρειαζόμαστε τη στήριξη και τη στήριξη των ομάδων μας οι οποίοι ε, κάνουν τεράστια προσπάθεια ώστε να μπορέσουν να προλάβουν όλες αυτές τις αποφάσεις από τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να διοχετεύσουν τις ε, ενισχύσεις ε, στις επιχειρήσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την υποστήριξη και για την αναγνώριση ε, της δουλειάς που κάνουμε 7 μέρες ε, την εβδομάδα, 24 ώρες το 24ωρο, ώστε να είμαστε στο πλευρό των κρατών μελών, ώστε να μπορέσουμε να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις σε μια αυτή την κατάσταση η οποία είναι άνευ προηγουμένου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Ευχαριστούμε κυρία Βεστάγκερ για την ε, συνεργασία σας και απομείνατε περισσότερο από ό,τι προβλεπόταν. Είδατε ότι είναι πολλές οι ερωτήσεις και πολύ το ενδιαφέρον για όσα κάνετε. Βεβαίως θα είμαστε σε επαφή. Και βεβαίω για την επερχόμενη έκθεση για τον ανταγωνισμό που πρέπει να συζητήσουμε σίγουρα τον Ιούνιο. Θα έχουμε και άλλες ευκαιρίες σύντομα για να το συζητήσουμε. Ευχαριστώ και τους ε, διερμηνείς και όσους το κάνουν εφικτό όλο αυτό, παρά τις δυσμενείς συνθήκες. Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε όλους. Ε, λίγη